Καλημέρα σας. Ε, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη συνεδρίαση της υποεπιτροπής μας. Υπάρχει διερμηνία στις εξής γλώσσες. Γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, εστονικά, ουγγρικά, λιθωνιακά, πορτογαλικά και ρουμάνικα. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις επί του σχεδίου της ημερησίας διάταξης, θεωρείται ότι έχει υιοθετηθεί. Πάμε τώρα στι ανακοινώσει του Προέδρου. Αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρου του Προέδρου, τη Προέδρου, κυρία Λουαζό, θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι σε συνέχεια τη πρόσκληση από τον κύριο Mr. George Ντόμερκ, Γενικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα, η επίσκεψη εργασία τη Επιτροπή μα θα λάβει χώρα στι 18 Νοεμβρίου από τι 12 μέχρι τι 2 η ώρα το μεσημέρι, έχοντα υπόψη προηγούμενε ανάλογε επισκέψει μέχρι 15 μέλη της Επιτροπής θα μπορούν να συμμετάσχουν. Η Γραμματεία της Επιτροπής είναι υπεύθυνη για την οργάνωση της επίσκεψης εργασίας σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του οργανισμού. Λόγω της συμμετοχής της κυρίας Λουαζό στη συνεδρίαση για την αξιολόγηση της ακρόασης του υποψηφίου για την θέση του ΥΠΑΤΟ εκπροσώπου και αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μπορέλ, τη συνεδρίαση, συνεδρίαση θα προεδρεύσουμε οι δύο αντιπρόεδροι Επιτροπής. Ας μην χρονοτροβούμε τώρα άλλο, καθώς η μερσία ατζέντα έχει αρκετά και ενδιαφέροντα ζητήματα. Ξεκινάμε με την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση και τις προοπτικές του έργου της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας. Θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω τους ομιλητές μας. Τον κύριο Άρνουτ Μόλναρμ, προϊστάμενο του Τμήματος Αμυντικής Πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ένωσης, τον κύριο Φρανκ Ντέζι, αναπηρωτή Διευθυντή Δυνατοτήτων Εξοπλισμού και Σχεδιασμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και τον Χρήστο Λαμπρόπουλο, συνταγματάρχη, μέλος του στρατιωτικού προσωπικού της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Τον Δεκέμβριο του 2017, 25 χώρες αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν το άρθρο 42 παράγραφο 6 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ξεκινήσουν τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία έχοντας ένα κεφάλαιο στην Ευρωπαϊκή Άμενα και να ενισχύσουν έτσι την αμυντική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΠΕΣΚΟ, όπως είναι γνωστή, αποτελεί το πολιτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη μεταξύ άλλων κοινών εξοπλιστικών και επιχειρησιακών προγραμμάτων. Με την ένταξή τους τα κράτη-μέλη ανέλαβαν οικονομικές και άλλες δεσμεύσεις για την περαιτέρω εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων οι δεσμεύσει αυτέ αντανακλούν τη φιλοδοξία για μια Ευρώπη που θα μπορεί να ανταπεξέλθει στι σύγχρονε προκλήσει και να μπορεί να προστατέψει έτσι αποτελεσματικά του πολίτε τη. 34 προγράμματα έχουν ήδη μπει κάτω από την ομπρέλα τη ΠΕΣΚΟ και ένα ακόμα ετοιμάζεται να εγκριθεί από το Συμβούλιο. Α ακούσουμε όμω του ομιλητέ μα. Κύριε Μόλεναρ, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Μετά είναι ο κύριο Δέζιτ και τελευταίο ο κύριο Λαμπρόπουλο. Thank you very much. Uh, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση για να σας παρουσιάσουμε πώς έχουν τα πράγματα με την ΠΕΣΚΟ. που τότε που ξεκίνησε, το Δεκέμβριο του 2017, γίνει πολλή δουλειά σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Πριν επανέλθω στα τρέχοντα θέματα, να κάνουμε μια επισκόπηση, να θέσω το πλαίσιο. Όπως ξέρετε, η μόνιμη διαθρωμένη συνεργασία προβλέπεται στην ε, Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενεργοποιήθηκε το 2017 με βάση τη στρατηγική της Ένωσης και το γενικότερο πλαίσιο του 2016. Το Συμβούλιο αποφάσισε να διερευνήσει τις δυνατότητές του. Στο τέλος του 2017, σε μια κοινή ανακοίνωση προς το Συμβούλιο, 25 κράτη-μέλη ανέλαβαν 20 δεσμεύσεις μεταξύ τους στους πέντε τομείς που αναφέρει το πρωτόκολλο της ΠΕΣΚΟ, το οποίο είναι παράρτημα των συνθήκων. Σε αυτή τη βάση το Συμβούλιο πήρε την απόφαση να δημιουργηθεί η ΠΕΣΚΟ. Μερικά βασικά σημεία διακυβέρνηση τη ΠΕΣΚΟ, οι αποφάσει και συστάσεις από το Συμβούλιο στα πλαίσια τη ΠΕΣΚΟ λαμβάνονται μέσω ψηφοφορία των συμμετεχόντων κρατών μόνο. Συμμετέχουν και τα 28 κρατη κατά τις συζητήσεις για την ΠΕΣΚΟ, αλλά οι αποφάσει λαμβάνονται μέσω ψηφοφορία των 25 μόνο. Τα κράτη-μέλη, αυτά τα 25, είναι ατομικά υπεύθυνα και λογοδοτούν για να ε, εκπληρώσουν τις πιο δεσμευτικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. Γι' αυτό έχουν εθνικά σχέδια εφαρμογής, τα οποία υποβάλλονται στην αρχή κάθε χρόνου για να είναι η βάση για την διαδικασία αξιολόγησης που ε, έχει δημιουργηθεί. Τρίτον, τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν συμμετέχουν και σε κοινά προγράμματα για να εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους. Δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη σε όλα τα προγράμματα και ε, βεβαίως στα προγράμματα αυτά δεν συμμετέχουν άλλοι που δεν είναι μέλη της ΠΕΣΚΟ, αλλά γίνεται ετήσια αξιολόγηση. Επίσης έχουμε μια διαδικασία για να εξεταστούν τα νέα προγράμματα που κατόπιν εγκρίνονται από το Συμβούλιο. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα για τρίτη φορά ε, επί του παρόντος. Η γραμματεία της ΠΕΣΚΟ αποτελείται από την Υπηρεσία Κοινή Δράσης, την ΣΕΚ και το στρατιωτικό προσωπικό και την, ε, το φορέα άμυνα. Συνεργαζόμαστε με συντονισμένο τρόπο. Είναι ένα ενιαίο σημείο επαφής για τα κράτη-μέλη και έχουμε και ένα κοινό ηλεκτρονικό χώρο εργασία. Πέμπτον, ο ύπατος εκπρόσωπος είναι υπεύθυνο για την ετήσια έκθεση που γίνεται στο Συμβούλιο για την ΠΕΣΚΟ για να εξετάσει πώ εφαρμόζει η ΠΕΣΚΟ τα προγράμματά τη και αναφέρεται και ο βαθμό εκπλήρωση των δεσμεύσεων κάθε κράτου μέλου. Η πρώτη ετήσια έκθεση δημοσιεύθηκε τον περασμένο Μάρτιο. Επίση, στέλνουμε και συστάσει προ το Συμβούλιο όσον αφορά τις προτάσεις προγραμμάτων. Όπως σας είπα αυτή η διαδικασία είναι να εξελίξει αυτή τη στιγμή με τον, αντιπρόεδρο και τον επικεφαλής του Οργανισμού Άμυνας προσπαθούμε να υπάρχει συνέπεια στην εφαρμογή όλων των πρωτοβουλειών άμυνας, όχι μόνο της ΠΕΣΚΟ, αλλά σχετίζεται και με την ετήσια συντονισμένη επισκόπηση της άμυνας, το ΚΑΡΔ, και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Το βασικό είναι να χρησιμοποιήσουμε τις 11 προτεραιότητες ανάπτυξης δυνατοτήτων της Ένωσης που συμφωνήθηκε όταν δημιουργήθηκε ο Οργανισμός Άμυνας. Αυτή είναι η βάση και για το ΚΑΡΤ και για το Ταμείο της Άμυνας. Εδώ βλέπουμε για παράδειγμα πού μπορεί να υπάρξει πρόβλημα για να το αντιμετωπίσουμε. Η Επιτροπή δεν έχει απευθείας ρόλο στη διακυβέρνηση της ΠΕΣΚΟ, αλλά είναι συνδεδεμένη με τις διαδικασίες στο Συμβούλιο και μπορεί να προσκληθεί για να συμμετάσχει και στις διαδικασίες κάποιων προγραμμάτων της ΠΕΣΚΟ για να υπάρχει συνεργασία με οργανισμούς ε, των οποίων ηγείται η Κομισιόν, όπως για παράδειγμα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας. Τι έχουμε κάνει λοιπόν από το που ξεκίνησε η ΠΕΣΚΟ. Πρώτα απ' όλα συμμετέχουμε με, με τα κράτη-μέλη στη διαδικασία καθορισμού των στόχων. Για παράδειγμα το Συμβούλιο ενέκρινε γενικού κανόνε διακυβέρνηση για τα προγράμματά μα, ούτω ώστε όλα τα προγράμματα να ακολουθούν ε, του ίδιου γενικού κανόνε. Δεύτερο, το Συμβούλιο καθόρισε και πιο ακριβεί στόχου για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων τη ΠΕΣΚΟ, ούτω ώστε να είναι ο οδηγό για την ε, εκπόνηση των εθνικών προγραμμάτων εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Και πρόσφατα έχουμε και μια απόφαση του Συμβουλίου με τις γενικές συνθήκες μέσω των οποίων και Τρίτε χώρες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε προγράμματα της ΠΕΣΚΟ. Έχει υπάρξει ουσιώδη πρόοδος για το θέμα αυτό, παρά την περιπλοκότητα του θέματος. Διότι τα προγράμματα της ΠΕΣΚΟ είναι βεβαίως ε, ουσιοδό ε, προγράμματα της Ένωσης. Και αυτό οδηγεί σε συγκεκριμένες συνθήκες τις οποίες θα πρέπει να πληρούν όσα κράτη, όσα, όσες τρίτες χώρες θέλουν να συμμετάσχουν. Η Φιλανδική Προεδρία θα πρέπει να ολοκληρώσει αυτή την προσπάθεια. Επίση, έχουμε ξεκινήσει 34 προγράμματα τη ΠΕΣΚΟ και μία τρίτη δέσμη εξετάζεται αυτή τη στιγμή από τα κράτη-μέλη για να εγκριθεί από το Συμβούλιο το Νοέμβριο. Έχουμε και κάποια κριτήρια αξιολόγηση για να εξετάσουμε τα νέα αυτά προγράμματα. Να αξιολογήσουμε καθώ θα πρέπει να εφαρμοστούν. Υπάρχουν αρκετά προγράμματα ήδη. Το Eurodrone, η Ευρωπαϊκή Δίκηση για ιατρικά θέματα για να αντιμετωπίσουμε επίσης διάφορα κενά που εντοπίστηκαν από την αξιολόγηση των δυνατοτήτων. Επίσης, για πρώτη φορά, λάβαμε τεχνικά προγράμματα εφαρμογής και κάναμε μια τεχνική αξιολόγηση αυτών των NIP, όπως θα αποκαλούμε, από τη γραμματεία της ΠΕΣΚΟ και αυτό κατέληξε στην ετήσια έκθεση της ε, υπάτης εκπροσώπου προς το Συμβούλιο που δεν είναι δημόσιο όμως γιατί διάφορα που περιέχουν ε, δια, ε, διαβαθμισμένη προφόρηση. Αλλά υπήρξε και μία δημόσια ανακοίνωση για να, καθαρίσουμε, να καθορίσουμε τα κριτήρια εφαρμογή από τα κράτη-μέλη των προγραμμάτων μας. Ορισμένα κράτη-μέλη σημείωσαν ότι υπάρχει αύξηση των εθνικών προπολογισμών άμυνα. Είναι μία από τι πρώτε δεσμεύσει τη ΠΕΣΚΟ και για τον τομέα των κοινών επενδύσεων για την άμυνα. Χρειάζεται περισσότερη εργασία, ούτω ώστε οι επενδύσει αυτέ να ενισχύσουν την ε, συλλογική ανάπτυξη δυνατοτήτων και τι ε, δυνάμει που χρησιμοποιούμε στι διάφορε αποστολέ. Από τα 34 προγράμματα το Συμβούλιο είπε έγιναν πολλά καλά αλλά κυρίως πρέπει να γίνουν περισσότερα για την εφαρμογή. Επίσης, το 2020 το Συμβούλιο αποφάσισε να μην υπάρξουν νέα προγράμματα. Το 2020 δηλαδή θα εφαρμόσουμε τα υπάρχοντα και τα νέα προγράμματα θα υπάρξουν το 2021. Πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα και η λεπτομέρεια των στοιχείων που υπάρχουν στα ΝΥΠ και επίσης είπαμε ότι πρέπει να προετοιμάσουμε το έδαφος για τη στρατηγική αξιολόγηση της ΠΕΣΚΟ που θα γίνει το 2020. Αυτή η αξιολόγηση, η αναθεώρηση είναι ακόμη νωρί, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη συζητήσει με τα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την ε, εφαρμογή των κριτηρίων και την ε, συνέπεια. Επίσης, η εκπρόσωπος ανέλαβε δέσμευση για κάποιες νέες ιδέες που θα υποβληθούν τον επόμενο Μάρτιο-Απρίλιο, αλλά πρέπει να γίνουν και περαιτέρω συζητήσεις με τα κράτη-μέλη για το περιεχόμενο αυτών των νέων συστάσεων και το, και το πεδίο εφαρμογή. Και με χαρά θα ενημερώνουμε τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί η πολιτική σας στήριξη είναι πολύ σημαντική, ούτως ώστε να υπάρχει συνέπεια και συνεκτική λογική στην όλη προσπάθεια. Έχουμε με όλα αυτά τα μέσα την ευκαιρία η ευρωπαϊκή άμυνα να αλλάξει πορεία ριζικά. Η συνεργασία να είναι το σύνηθες. Να επενδύουμε περισσότερα και από κοινού για τις σωστέ δυνατότητες και τη σωστή χρήση και τη συντονισμένη χρήση. Έτσι θα ενισχύσουμε τη στρατηγική μας αυτονομία και θα ωφεληθεί και το ΝΑΤΟ και σα ευχαριστώ πολύ. Διακεκριμένα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε καταρχά για την πρόσκλησή σα να έρθω και να μιλήσω στην Επιτροπή Άμυνα και Ασφαλεία. Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σα σήμερα και έχω τη δυνατότητα να σα ενημερώσω για την ΠΕΣΚΟ. Κάνοντα το αυτό, θα εστιαστώ στι δραστηριότητε ίδιε και τι δραστηριότητε εντό γραμματεία τη ΠΕΣΚΟ. Καταρχά, θα ήθελα να βασιστώ σε αυτά που είπε η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση θα πρέπει να κάνουμε επισκόπηση της ΠΕΣΚΟ στα πλαίσια τη υπηρεσία εξωτερική δράση για την υποστήριξη των κρατών μελών στι προσπάθειε να αυξήσουν τι δυνατότητέ του με έναν τρόπο συνεργατικό. Η Παγκόσμια Στρατηγική για ΚΕΠΑ και σχετικέ δραστηριότητε ε, αφορά στενότερη στενοργασία όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια. Ταυτόχρονα, ανοίξαμε το δρόμο για σειρά πρωτοβουλειών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και θέλουμε να ενισχύσουμε τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά σχεδιασμό να αναθεωρήσουμε τη, τα σχέδια ανάπτυξης δυνατοτήτων CDP. Θέλουμε συντονισμένη ετήσια ε, έκθεση, την CARD για την άμυνα και να δημιουργηθεί και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το EDF. Το CARD, το EDF και η PESCO είναι αλληλένδετα και δρομολογούν διάφορες πρωτοβουλίες με έναν απλουστευμένο τρόπο. Μπορούμε να πούμε ότι αναθεωρημένη το σχέδιο δημιουργίας δυνατοτήτων και το, οι αναπτυξιακέ προτεραιότητε για το 2018 τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω μα λένε πού πρέπει να εστιάσουμε τι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Η συντονισμένη ετήσια έκθεση για την άμυνα μα δίνει μια γενική εικόνα του πού βρισκόμαστε, εντοπίζονται τα επόμενα βήματα και ανοίγει το δρόμο για νέα ε, προσπάθεια συνεργασία σε διάφορου τομεί, συμπεριλαμβανομένου τη ΠΕΣΚΟ. Η ΠΕΣΚΟ μα δίνει επιλογέ. Πώ μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μέσω συνεργασία και διαθρωμένα και έχουμε ένα πλαίσιο για να μπορούμε να σχεδιάζουμε όλοι μαζί. Και το EDF θα δώσει επίσης τα χρήματα για την άμυνα, τα κοινά προγράμματα, του Ευρωπαϊκού Τομείο Άμυνας, το EDF, ε, εντός της ε, ΠΕΣΚΟ. Σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι πρωτοβουλίες συντονίζονται ομαλά. Υπάρχει τέλειος συγχρονισμός. Είναι ένα κομμάτι των στόχων. Έχουν δεσμευτεί τα κράτη-μέλη να τα εφαρμόσουν αυτά ε, μέσω εφαρμοστικών σχεδίων τα κράτη-μέλη στα πέσχα της ΠΕΣΚΟ και κάνουμε προσπάθεια να κινηθούμε έτσι στην ΠΕΣΚΟ όταν αξιολογούμε τα διάφορα προγράμματα. Τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειε του συστήματος διαχείρισης. Υπάρχουν δύο στιβάδες. Σε επίπεδο Συμβουλίου εξετάζουμε την κατεύθυνση που ακολουθούμε και λαμβάνονται οι αποφάσεις, γίνεται αξιολόγηση κατά πόσο τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν ανταποκρίνουν τι υποχρεώσει τους και δεύτερον σε επίπεδο διαχείριση προγραμμάτων και εκεί συμμετέχουν τα διάφορα κράτη-μέλη στα διάφορα προγράμματα της ΠΕΣΚΟ. Η γραμματεία της ΠΕΣΚΟ που αποτελείται από το ίδιο από τη μία πλευρά και από το Η EMS από την άλλη πλευρά θα υποστηρίξει την όλη προσπάθεια. Υποστηρίζει την όλη προσπάθεια. Η γραμματεία της ΠΕΣΚΟ συμβάλλει στην ετήσια έκθεση της ΥΠΑ εκπροσώπου για την ΠΕΣΚΟ, συντονίζει την αξιολόγηση των προτάσεων για προγράμματα των κρατών μελών, καθώς και κάνει αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων υλοποίησης για να δούμε κατά πόσο επιτυγχάνονται οι συμπεφωνημένοι στόχοι από πλευρά μελών. Πέραν αυτών, η γραμματεία τη ΠΕΣΚΟ ιχνηλατεί την πρόοδο σε αυτά τα προγράμματα τη ΠΕΣΚΟ και παρέχει βοήθεια στα κράτη-μέλη σε όλε τι πτυχέ τη αξιολόγηση και τη υλοποίηση τη ΠΕΣΚΟ. Η EDA, σαν τμήμα τη γραμματεία ΠΕΣΚΟ, έχει και άλλο ειδικό ρόλο να αποφύγει αλληλεπικάλυψη προσπαθειών και να διευκολύνει την ανάπτυξη δυνατοτήτων και των σχετικών προγραμμάτων άξιων Τώρα, πού βρισκόμαστε. Μέχρι τώρα, 25 κράτη τη Ευρωπαϊκής έχουν ενταχθεί στην ΠΕΣΚΟ και προσπαθούν να αποκριθούν στι υποχρεώσει μέσω επενδύσεως, σχεδιασμού, αναπτύξεως, δυνατοτήτων άμυνας εντός του πλαισίου τη Ευρωπαϊκής Ενώσεω. 34 προγράμματα ΠΕΣΚΟ έχουν επιλεγεί μέχρι τώρα και καλύπτουν 7 τομεί εκπαίδευση, κατάρτιση, ενημέρωση και συστήματα, αεροπορικά συστήματα, θαλάσσια συστήματα, ε, διαστημικά συστήματα, ε, κυβερνοσυστήματα και κοινέ ε, προσπάθειες χρήσης των πόρων. 17 προγράμματα θετήθηκαν από το Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2018. Δεύτερη φάση 17 άλλων προγραμμάτων τον Νοέμβριο του 2018 ενεκρίθησαν Άλλη μια ομάδα προτάσεων προγραμμάτων ΠΕΣΚΟ έχει δρομολογηθεί, έχει αξιολογη, έχουν αξιολογηθεί και επιλογή των προτάσεων αναμένεται να εθετηθεί τον Νοέμβριο φέτος. Μέσα, ο συνολικός αριθμός λοιπόν των προγραμμάτων πιθανότατα θα φτάσει περίπου στα 50 προγράμματα, θα καλύψουμε όλους τους τομείς ε, δυνατοτήτων αμυντικών. Σημασία έχει βέβαια η ποιότητα και όχι η ποσότητα και έχουμε αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο προγραμμάτων. Θέλουμε να είναι στέρεο το πλαίσιο, να είναι καλή βάση για την επιτυχία της ΠΕΣΚΟ και να εμπλουτίζουμε την, ε, τους στόχους που θέτουμε. Κάθε πρόγραμμα υλοποιείται από διάφορες ομάδες ε, μελών κρατών που συμμετέχουν στο ΠΕΣΚΟ και υπάρχει συντονισμός από ένα ή περισσότερα κάτι μέλη ε, πέσκο, των κρατών μελών της ΠΕΣΚΟ με συντονιστών. Μπορεί να συμφωνήσουν τα μέλη της ΠΕΣΚΟ όσον αφορά τη συμμετοχή των κρατών μελών ΠΕΣΚΟ, ποια, να συμμετέχουν και ποια κράτη θα είναι παρατηρητές σε ένα πρόγραμμα. Δεν θα εκπλήσει κανέναν ότι όπως υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις, υπάρχει και διαδικασία για την παραγωγή προγραμμάτων ΠΕΣΚΟ και πρέπει να υπογραμμίσω ότι είναι αυστηρή διαδικασία με πλήρη ε, κριτήρια αξιολογήσεως. Πώς λειτουργούν αυτά στην πράξη η διαδικασία ξεκινά με προκήρυξη διαγωνισμού για υποβολή προτάσεων από τη Γραμματεία. Παραλαμβάνονται οι προτάσεις, αξιολογούνται από τη Γραμματεία της ΠΕΣΚΟ. Οι προπτικές δυνατοτήτων αξιολογείται από την ΔΙΕ εφαρμόζοντας κριτήρια όπως είναι η συνοχή ε, του τοπίου των δυνατοτήτων, η οριμότητα των προτάσεων, συνοχή ε, κατά πώς συνάδουν με τις επιταγές του ΝΑΤΟ και οικονομική υποστήριξη. Σημαίνει ότι αξιολογούμε κατά πόσο ήδη ε, συμμορφώνονται τι απαιτήσει περεναρμόνιση που είναι κάτι απαραίτητο ξεκινήσει συνεργασία ή αν υπάρχει οδικό χάρτη για την εναρμόνιση. Επίση, εξετάζουμε και το επίπεδο συνοχή με τι δρομολογηθήσει δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Προσπαθούμε να βρούμε συνέργειε και πώ συνάδουν όλα αυτά με τι δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για να αποφύγουμε επικαλύψει των προσπαθειών και πολλαπλασιασμό των προσπαθειών και εξετάσουμε ενδεχόμενε δυνατότητες επιχειρηματικές, ανάλυση κόστους κόστους-οφέλους των διαφόρων προγραμμάτων. Η επιχειρησιακή αυτή εικόνα αξιολογείται από την EUMS και βλέπουμε πώς οι προτάσεις γεφυρώνουν ενδεχόμενα κενά και ποια είναι τα ωφέλη που απορρέουν την υλοποίηση των προγραμμάτων. Τα κράτη-μέλη συμμετέχουν πλήρω εντό τη διαδικασία και από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η διαδικασία παρέχουν διευκρινήσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες για τη βελτίωση του συστήματος και υποστηρίζονται τα προγράμματά τους από άλλη κάτι μέλη μέσω της διαδικασίας έγκρισης των προτάσεων μέσω του Συμβουλίου της ΠΕΣΚΟ. Από τη στιγμή που ένα πρόγραμμα έχει συμφωνηθεί, το ο μέλος που έχει το συντονισμό του προγράμματος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από την ΕΔΗ για υποστήριξη πέρα από τα καθήκοντα της γραμματής ΠΕΣΚΟ. Μέχρι τώρα τέσσερα προγράμματα έχουν ε, τύχη υποστήριξη για τη θαλάσσια, μη αυτόνομα ε, συστήματα για την αρκαλίευση, το, για τα διφωνικά συστήματα, ταχύ ανταπόκριση για κυβερνοεπιθέσεις και βοήθεια για την κυβερνοασφάλεια και CBRNN εποπτείασαν ε, υπηρεσία. Για το τελευταίο πρέπει να πούμε ότι μια απόφαση ελήφθηκε από το συντονιστή του προγράμματος για να εφαρμοστεί αυτό σαν ένα EDA πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας πλήρως τα φελη που προέχει, παρέχει το πλαίσιο EDF ε, μέσω των διαφόρων εξαιρέσεων. Και ίσως και στο μέλλον να ακολουθήσουν και άλλα παραπρογράμματα. Τώρα να πω μερικά πράγματα για τα εθνικά σχέδια υλοποίησεως προγραμμάτων, κάτι που ανέφερα ήδη. Η σύσταση του Συμβουλίου αφορά την, τη σειρά που θα ακολουθούν θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που έχουν αληφθεί στα πλαίσια τη ΠΕΣΚΟ με πιο ακριβείς στόχους που καθορίζονται και απαιτείται από τα κάτι μελη να μοιράζονται μία φορά το χρόνο τα εθνικά εφαρμοστικά σχέδια για να δείξουν σε ποιο επίπεδο έχουν πετύχει και έχουν υλοποιήσει τις υποχρέωσεις που έχουν αναλάβει στα πλαίσια της ΠΕΣΚΟ. Η γραμματεία της ΠΕΣΚΟ θα πρέπει να αξιολογήσει τα εθνικά εφαρμοστικά σχέδια από πλευράς δημιουργία δυνατοτήτων υπό την ευθύνη τη CDA και τα επιχειρησιακά στοιχεία που είναι ευθύνη τη υπηρεσίας εξωτερική δράση. Η ετήσια έκθεση για την ΠΕΣΚΟ εδράζεται επί της τροφοδοσίας πληροφοριών τη γραμματεία του ΠΕΣΚΟ και δίδεται, θα δοθεί το Μάρτιο 2020 στο Συμβούλιο για να γίνει η περιστατωμένη συζήτηση για την υλοποίηση του ΠΕΣΚΟ στα πλαίσια του, από πλευρά των κρατών μελών. Η γραμματεία του ΠΕΣΚΟ διευκολύνει την όλη διαδικασία και υποστηρίζει τα κράτη-μέλη για να προωθήσουν τους διάφορους στόχους. Τώρα που μιλάμε, ένας δεύτερος γύρος διμερών συνομιλιών με τα κράτη-μέλη λαμβάνει χώρα και τα κράτη-μέλη την χάνουν υποστηρίξεω για να βελτιώσουν καλύτερα την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους και να ολοκληρώσουν τις πληροφορίες που παρέχουν. Ε, τα διάφορα έγγραφα, εργαστήρια, βοήθεια είναι συμπληρωματικά στοιχεία τη όλη αυτή διαδικασία, Όλα αυτά μαζί αποτελούν ένα τμήμα τη καθημερινή μα δουλειά που κάνουμε για να υποστηρίξουμε την υλοποίηση των σχεδίων ΠΕΣΚΟ και βοηθούμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ΠΕΣΚΟ για το μέλλον της Ευρώπης. Τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό, βάσει αυτών των αρχικών εμπειριών των δραστηριοτήτων που αφορούν τα προγράμματα και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλυφθεί, το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του τη 19 η Νοεμβρίου του 2018 κάλεσε τη γραμματεία τη ΠΕΣΚΟ να παρουσιάσει μια έκθεση όσον αφορά την αρχική επιτυχία των προγραμμάτων έκανε αυτή την έκθεση, το υπέσκο σε στενή ε, συνεργασία με τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη και μέσω του εγχειρήματο διαφάνει ότι κάποια συμμετέχοντα κράτη-μέλη ήταν υπέρ του να εστιαστούμε το να χορηγούν τα αποτελέσματα των προγραμμάτων της ΠΕΣΚΟ αντί να αναπτύσσουν νέα προγράμματα. Δηλαδή να δούμε τι γίνεται με αυτά που ήδη έχουν δρομολογηθεί. Και έχουμε τον πρώτο κύκλο των CARD που θα οδηγήσει σε μια έκθεση τον Νοέμβριο του 2020 έχοντας την, τη νέα κλίση για υποβολή προτάσεων ε, το 2021 μόλις. Τα αποτελέσματα των ΚΑΡΤ μπορούν να τα εκμεταλλευτούμε να το εκμεταλλευτούν τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν για να δουν νέους δρόμους για τη διαδικασία. Δεν προβλέπεται άλλη υποβολή προτάσεων τον επόμενο χρόνο και αυτό είναι το πρώτο σημαντικό βήμα προσπάθεια συντονισμού CARD και PESCO. Η σύσταση του Συμβουλίου ανοίγει οδικό χάρτη για την υλοποίηση των προγραμμάτων μέσω στρατηγική αναθεώρηση ΠΕΣΚΟ στο τέλος πρώτη φάση, τη πρώτη διετία, για να αξιολογηθεί κατά πόσο εκπληρωθεί η δεσμεύση τη ΠΕΣΚΟ. Αυτή η στρατηγική αναθεώρηση προβλέπεται, αυτή η έκθεση προβλέπεται αρχές του 2020 και θα δώσει κάποιε κατευθύνσει για τα 34 προγράμματα που θα δρομολογηθεί. Εδώ κλείνω αυτή την εισαγωγή και σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ο Λαμπρόπουλο. Σα eh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε από τα μέλη της Επιτροπής Άμυνα, με την παρέμβασή μου. Θα ήθελα να σας δώσω μια γενική εικόνα των ενεργειών που έχουν αναλάβει ε, ως μέλη της ε, γραμματείας ε, ΠΕΣΚΟ, το στρατιωτικό προσωπικό, καθώς επίση και τη χρήση που κάνουμε των επιχειρησιακών σχεδίων των εθνικών, όπως ήδη είπαν οι συνάδελφοι. Το στρατιωτικό προσωπικό λειτουργεί ως στο πλαίσιο της γραμματείας ε, ΠΕΣΚΟ, στο πλαίσιο του, όπως περιγράφεται στο άρθρο 7, της απόφασης 2315 του Συμβουλίου του 2017 και πιο συγκεκριμένα συνεισφέρουν στην επιχείρηση, στα... Ε, στα επιχειρησιακά και στην αξιολόγηση που γίνεται ετησίως. Επίσης, στον συντονισμό ε, έργων ιδίως όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και τη διαλειτουργικότητα των ε, δυνάμεων. Επίσης συνεισφέρουν επιχειρησιακά όπου χρειάζεται και θα επανέλθω πιο συγκεκριμένα σε αυτό. Επίσης, για την Στρατιωτική Επιτροπή, η UMS ε, προετοιμάζει την έκθεση η οποία Στρατιωτική Επιτροπή υποβάλλει στην Πολιτική Επιτροπή, με την οποία γίνεται η αξιολόγηση των προγραμμάτων ΠΕΣΚΟ, καθώς επίσης και μια αιτήσια έκθεση της εφαρμογής των προγραμμάτων ΠΕΣΚΟ. Η ΙΟΓΕΜΕΣ λοιπόν λειτουργεί και, στο πλαίσιο, και παρέχει αξιολόγηση λαμβάνοντας ε, συνεισφορές από όλες τις διευθύνσεις της EUMS και τους αντίστοιχους εμπειρογνώμονες. Αυτή η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται προκειμένου να εντοπισθούν ε, ε, στοιχεία που μπορεί να λείπουν και πρώτα απ' όλα επιδιώκουμε να τηρούμε τους κανόνες και τις διαδικασίες και τους αντίστοιχους στόχους ε, υψηλής προτεραιότητας. Ε, αυτή τη στιγμή έχει εντοπιστεί ένα project το οποίο μπορεί να συνεισφέρει στην ε, διαθεσιμότητα και διαλειτουργικότητα των δυνάμεων, δηλαδή τη δυνατότητά μας να συνεργαζόμαστε και να έχουμε κοινέ διαδικασίες. Αφού λοιπόν βρεθεί ένα project το οποίο μπορεί να συνεισφέρει προς αυτό, εξετάζουμε πώς μπορεί να συνεισφέρει στις στρατιωτικές φιλοδοξίες στο, στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα, στην, όπως σας είπα, διαθεσιμότητα και διαλειτουργικότητα των δυνάμεων. Έχουμε μια διαδικασία βάσει της οποίας αντλούμε διδάγματα και μετά από αυτή την προσπάθεια και μετά από αυτή την αξιολόγηση επιλέγονται τα προγράμματα ΠΕΣΚΟ τα οποία καλύπτουν πλήρως και τα, όλους τους κλάδους που καλύπτει η ΠΕΣΚΟ ε, είτε στις χερσαίες δυνάμεις, στις θαλάσσιες δυνάμεις, αέριες δυνάμεις, καθώς επίσης και κυβερνοσυστήματα και άλλα. Επίσης επιδιώκουμε άμεσα να καλύπτουμε κενά τα οποία μπορεί να έχουν εντοπιστεί σε επιχειρήσεις που διεξάγονται καθώς επίσης και να καλύπτουμε κοινά έτσι ώστε στο μέλλον να μπορούμε να καλύπτουμε το πλήρες φάσμα των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτή τη ε, διαδικασία αξιολόγηση, θα γνωρίζετε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει ετησίω να αναθεωρούν τα ετήσια ε, σχέδια υλοποίηση μέχρι τι 10 Ιανουαρίου συνήθω. Αυτή η διαδικασία στην οποία συμμετέχει και το ε, στρατιωτικό προσωπικό ε, πληρεί πλήρω τι τις που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο εφαρμόζονται τα κριτήρια για την ε, λεγόμενη περιοχή C, δηλαδή πώς μπορεί να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα και η λειτουργικότητα των δυνάμεων, εντοπίζοντας κοινού στόχους. Και αυτό πιθανώς να οδηγήσει σε επαναξιολόγηση εθνικών αποφάσεων τα κράτη-μέλη τα οποία αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της, του τομέα C ε, κάποιες δεσμεύσεις, αξιολογούν τα επιτεύγματά τους και κάνουν προβολές, ε, κάποιες προβλέψεις μάλλον, για, ε, βραχυπρόθεσμα για τον επόμενο χρόνο και πιο μεσοπρόθεσμα για τα επόμενα πέντε χρόνια. Με αυτές τις πληροφορίες αξιολογείται κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε τις δύο προτεραιότητες 13, για τη διαλειτουργικότητα, 14 για την ε, χρηματοδότηση των κοινών επιχειρήσεων και τις αντίστοιχες ε, δεσμεύσεις που πηγάζουν από αυτές. Όπως ε, έλεγα λοιπόν, το στρατιωτικό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί στο πλαίσιο της γραμματείας ΠΕΣΚΟ, προσπαθώντας να εξειδικεύσει τους γενικούς στόχους high capability, υψηλών υψηλής σε πιο συγκεκριμένα προγράμματα. Σας ευχαριστώ. Και ο λόγος τώρα στα μέλη μας για ερωτήσεις. Mr. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτή την ε, ολοκληρωμένη παρουσίαση και χρήσιμη επισκόπηση της κατάστασης και των προοπτικών της ΠΕΣΚΟ. Λοιπόν, να ζητήσω μερικές περαιτέρω επεξηγήσεις μέσω ερωτήσεων. Πρώτον, η ΠΕΣΚΟ είναι μια πολύ νέα δομή συνεργασίας και δεν έχει υπάρξει τόση εφαρμογή για να κάνουμε αξιολόγηση της κατάστασης. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες ε, δυσχέρειες. που να βοηθήσουν ούτως ώστε να είναι πιο αποτελεσματική ως επιχειρησιακή πλατφόρμα η ΠΕΣΚΟ στο μέλλον. Δεύτερον, η ΠΕΣΚΟ είναι σημαντική για να συνδυαστούν τα κράτη-μέλη και ήδη υπάρχει κάποια διαδικασία συντονισμού και θα πρέπει να συνεχιστεί το εκτιμώ ιδιαίτερα. Ελπίζω στο μέλλον να υπάρξουν 7 ε, τομείς συνεργασίας που θα μπορούσε να εμβαθυνθούν σε πιο ειδικευμένους τομείς για να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Ποια είναι όμως η σχέση μεταξύ ΠΕΣΚΟ και Ταμείου Άμυνας. Πώς θα αξιοποιήσετε το Ταμείο Άμυνας για να στηρίξετε, να χρηματοδοτήσετε ορισμένα προγράμματα ΠΕΣΚΟ. Και αν όχι, γιατί όχι. Και αν ναι, μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα. Και τρίτον, προτίθεστε να καλέσετε και τρίτα κράτη. Γιατί η ασφάλεια είναι ενιαία. Άρα χρειαζόμαστε να συνεργαστούμε με περισσότερους εταίρους από την γειτονία μας. Για παράδειγμα, εταίρους από επιχειρήσεις των οποίων ηγείται το ΝΑΤΟ. Και αν ε, σκοπεύετε να προσκαλέσετε να συμμετάσχουν και τρίτες χώρες με τι κριτήρια και έχετε κανένα παράδειγμα ήδη ή κάποιες προθέσεις συνεργασία στο μέλλον θα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα θα ήταν απόλυτα σωστό να συμμετάσχουν και τρίτες χώρες ως συνδεδεμένοι στα εγχειρήματα της ΠΕΣΚΟ. Good morning and thanks for your very... Καλημέρα σας. Πολύ ολοκληρωμένη παρουσίαση. Ευχαριστώ. Ε, πρώτη ερώτηση επιχειρησιακές δυνατότητες που προκύπτει από την ΠΕΣΚΟ. Τη φτιάξαμε την ΠΕΣΚΟ για να αυξηθεί η επιχειρηματική μας ε, ικανότητα. Έχουμε 34 προγράμματα. Τα περισσότερα όμως είναι έρευνα και ανάπτυξη. Για αυτή τη νέα δέσμη όμως θα υπάρξουν περισσότερα προγράμματα για δράση, για να ενισχύσουμε την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Και μετά η διαλειτουργικότητα. Η ΠΕΣΚΟ θέλει να αυξήσει και την ε, διαλειτουργικότητα από ό,τι καταλαβαίνω. Διαλειτουργικότητα των εθνικών ενόπλων δυνάμεων των διαφόρων κρατών μελών. Υπάρχουν προγράμματα για να καθορίσουμε με τεχνικούς όρους την διαλειτουργικότητα, για παράδειγμα πιστοποίηση, τυποποίηση, όχι μόνο για τις προδιαγραφές των κρατών μελών, αλλά και του ΝΑΤΟ και ανταλλαγή και υποβολή εκθέσεων μεταξύ κρατών μελών. Είπατε το CARD και τα NIP ...όσο καλά από πλευρά διαφάνεια, ακρίβεια και κατάλληλη χρονική στιγμή είναι, είναι, προχωρά αυτά τα σχέδια. Ευχαριστώ. Η ερώτησή μου είναι προς τον κύριο Ντεζίτ. Στόχος της πέσκο. είναι ο συγχρονισμός των ε, δομών των εθνικών ενόπλων δυνάμεων. Πριν από δύο χρόνια το Spiegel, ένα γερμανικό περιοδικό, είχε μια ενδιαφέρουσα έκθεση για την Πέσκο όπου έλεγε ότι η Πέσκο θα είναι ένα είδος στρατιωτικού Σέγγεν. Δηλαδή να προετοιμάσει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού. Οι προμήθειες της, ε, του γερμανικού στρατού είναι ένας ε, τεράστιος οργανισμός με πολύ εμπειρογνωμοσύνη αλλά παρόλα αυτά θεωρείται βράδυ κίνητος και αναποτελεσματικός. Υπάρχουν 27 ε, εθνικές υπηρεσίες στρατιωτικών προμηθειών στα 27 κρατη στα άλλα 27 κράτη-μέλη. Πώς προτίθεστε λοιπόν να βελτιώσετε ιδιαίτερα για τις προμήθειες και τους εξοπλισμούς, την έρευνα για τους εξοπλισμούς. Πώς προτίθεστε να συγχρονίσετε καλύτερα τις προσπάθειές μας μέσω της Πέσκου. Ευχαριστώ πολύ. Μπέργ και το λόγο έχει η κυρία Ντεμιρέλ. Η κυρία Ντεμιρέλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Άκουσα ότι ο απολογισμός των προσπαθειών της ΠΕΣΚΟ μέχρι τώρα δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικός και δεν έχουν προχωρήσει πολύ τα 34 προγράμματα. Και ορισμένα φαίνεται ότι θα σταματήσουν. Θα ήθελα να μάθω ποια έχετε σταματήσει. Επίσης, στις 30 Σεπτεμβρίου έμαθα ότι σχεδιάζονται 13 περαιτέρω προγράμματα και διαπιστώνω ότι πολλά από αυτά είναι μικρής διαστάσεων αλλά το Future Combat Air System, system και άλλα δεν αναφέρονται. Θα ήθελα να μάθω για ποιο λόγο. Υπάρχουν λόγοι. Μήπως έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτά τα μεγάλης διάστασης προγράμματα εξαρτώνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ή είναι εσωτερικές δυσχέρειες ή δεν βρίσκουμε επαρκείς εταίρους στην ΠΕΣΚΟ. Κάποιοι μπορεί να τα μπλοκάρουν. Θα με ενδιέφερε αυτό. Και κάτι προσωπικό. Περίεργο μου φαίνεται ότι ο κατάλογος των προγραμμάτων από ό,τι είδα στις 30 Σεπτεμβρίου δεν λάβαμε το κατάλογο αυτών των προγραμμάτων στο Brussels 2 στις 30 Σεπτεμβρίου. Θεωρώ ότι για λόγους διαφάνειας και κοινωνιστικού ελέγχου θα ήταν πολύ σκόπιμο να έχουμε το κατάλογο αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Γουάλα, ο λόγος σας. Ευχαριστώ πολύ. Διάφορα θέματα θέλω να θέσω για την Πέσκο. Στην Ιρλανδία υπάρχει διχογνωμία. Όταν ψηφίστηκε στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο, πολλοί από εμά ήμασταν αντίθετοι. Πέρασε όμω ο σχετικό νόμο. Αλλά μας ε, ανησυχεί κάπως η περαιτέρω στατικοποίηση της Ευρώπης δεν είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό είναι ο δρόμο για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Μιλήστε τη συνεργασία, ότι η φιλοδοξία πρέπει να ταιριάζει με του πόρου που διαθέτουμε. Και οι αμυντικέ μα δυνάμει ε, φεύγουν από τη χώρα μα. Φεύγουν οι άνθρωποι του στρατό γιατί δεν πληρώνονται. Και έχουμε και το θέμα του εξοπλισμού. Μπορεί να υπερβάλλουμε εκεί και να κοστίζουν πολλά χρήματα για νέο εξοπλισμό. θα μπορούσαν ίσως να αντικατασταθούν ε, με μοντέρνα μέσα που είναι πιο φθηνά, όπως με τα μη επανδρομένα ε, πτάμενα οχήματα, με τα drones. Το βλέπουμε, το κάνουν οι Σαουδάραβες. Έχουν αντιεροπορικό εξοπλισμό οι Σαουδάραβες θα μπορούσαν αντί να αγοράσουν τα πυραυλικά συστήματα εράμινα να βρουν την ίδια λύση με πιο φθηνά drones. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που μπορούμε να εξετάσουμε. Πολλές περιοχές έχουν αποσταθεροποιηθεί στη γειτονιά μας. Στο Ιρλανδικό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει μια έλλειψη συσχετισμού σκέψεων και προβληματισμού. Δεν κάνει αρκετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αντιμετωπίσει τους φορολογικούς παραδείσους. Αποσταθεροποιούμε, κλέβουμε πόρους από τις αναπτυσσόμενες χώρες, φεύγει ο κόσμος από την πατρίδα του και μεταναστεύει και πάει αλλού για να βρει δουλειά. Εάν θέλουμε να γίνει πιο ασφαλής η Ευρώπη, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους φορολογικούς παραδείσους και να μην παίρνουμε τους πόρους από τους ντόπιου ε, λαούς. Η χρήση κυρώσεων είναι σωστή. Άκουγα χθε τον κύριο Γιώσεφ Μπορέλ στην ακρόασή του. Είπε ότι δεν είναι υπερασπιστής των κυρώσεων Φεύγει ο κόσμο από τη Βενεζουέλα λόγω κυρώσεων. Δεν επιστρέφει ο κόσμο στη Συρία λόγω αυτού. Στον Περσικό κόλπο δημιουργήθηκε αποστεθαροποίηση. Δεν θα πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο να ανησυχούμε την ασφάλεια. Να μην χρησιμοποιούμε τόσο τις κυρώσεις, διότι είναι μια μορφή οικονομικής τρομοκρατίας οι οικονομικές κυρώσεις. Τα τελευταία χρόνια πολλές προσπάθειες που κάναμε στην Ευρώπη πολλοί, πολλές ε, στατιωτικές επεμβάσεις έγιναν να προστατευτούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην προσπάθεια εξόριξης ορυκτών όπως η Γαλλία ε, που κινήθηκε, δραστηριοποιήθηκε για αυτόν το σκοπό στο Μαλί. Λίγο πιο σύντομα. Ε, okay, I'll, I'll Καλώς, θα ολοκληρώσω σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μαυρίδης έχει το λόγο. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. I'm not the chair. Δεν είμαι εγώ πρόεδρος. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους τους ομιλητές μας. Έχω ένα διπλό ερώτημα. Δεν είμαι ούτε ειδικό στα στρατιωτικά, ούτε ειδικό σε τεχνικά θέματα. Εγώ συνεχίζω το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Μπέρκ. Αντιλαμβάνομαι ότι μέχρι τώρα, ή τέλος πάντων στο άμεσο μέλλον, η ΠΕΣΚΟ προβλέπεται να είναι ένας τρόπος οικονομικής συνεργασίας, να βρεθούν συνέργειες στα κράτη-μέλη που συμμετέχουν σε αυτή. Εγώ έχω μια περισσότερο πολιτική ερώτηση. Ποιος είναι ο βαθμός φιλοδοξίας για την ΠΕΣΚΟ στο μέλλον, δηλαδή πώς βλέπουμε να εξελίσσεται η ΠΕΣΚΟ στο μέλλον και κάτι ακόμα υπάρχουν πραγματικές απειλές, είτε αυτό μας αρέσει είτε όχι. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κράτος μέλος στην Κύπρο, η οποία προσπαθεί, της οποίας μάλλον η αποκλειστική οικονομική ζώνη ε, ε, παραβιάζεται από την Τουρκία. Τα, ε, τα ελληνικά σύνορα παραβιάζονται επίσης από την Τουρκία και αναφέρω μόνο αυτά. Υπάρχουν λοιπόν προτάσεις ή εργαλεία από την ΠΕΣΚΟ αυτή τη στιγμή να μπορούμε να αξιοποιήσουμε ή είναι μια συζήτηση που κάνουμε που κάποια στιγμή στο μέλλον θα τελεσφορεί. Ευχαριστώ. Έχει κάποιο άλλο συνάδελφο ερώτηση. Επί του θέματο όμω, όχι για του φορολογικού παραδείσου. Monsieur le Président, moi j'ai un point de procédure à soulever. Συγγνώμη. Αλλά όταν αρχίζει η συνεδρίαση τη υποεπιτροπή μα, έχουμε μια μερίσια διάταξη με θέματα τα οποία έχουν συμφωνηθεί και πρέπει να την ακολουθούμε. Αν αρχίζουμε να θέτουμε ερωτήσεις για οποιοδήποτε θέμα, επειδή απλώς έχουν γνώσεις για θέματα άμυνας ε, ή στρατιωτικών, θα πάμε προς κάθε κατεύθυνση. Κοιτάξτε, πρέπει να είναι οργανωμένες εργασίε μα. Θα μιλήσουμε βεβαίω κάποια στιγμή για την τρομοκρατία, θα μιλήσουμε για το Μαλί, αλλά τώρα συζητάμε για την Πέσκο. Έρχονται εδώ να μας μιλήσουν οι υπεύθυνοι του, της Πέσκο. Και βεβαίω μπορούμε να κάνουμε κάποιε διευρύνσει των ερωτήσεων, αλλά πρέπει να έχουν να κάνουν με την ουσία του θέματο. Θα σα ζητούσα κύριε Πρόεδρε να αξιοποιήσετε τι δυνατότητε που έχετε. Για να διακόπτετε τι παρεμβάσει που δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα που συζητάμε. Γιατί αλλιώς θα χρειαστούμε ώρες χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Γιατί οι ομιλητές μας δεν έχουν ερωτήσεις ε, και δεν αναμέναμε να έχουν ερωτήσεις για από τα θέματα που τους τίθενται. Σας παρακαλώ, εάν από την αρχή της θητείας μας δεν μάθουμε να λειτουργούμε σωστά, θα γίνουμε γελοί. Κανείς δεν θα έρχεται στην Επιτροπή μας, γιατί θα κάνουμε συζητήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την ημερήσια διάταξη η οποία έχει εγκριθεί. Σας παρακαλώ, λίγη πειθαρχία στην διεξαγωγή των εργασιών μας. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε κατά σειρά. Thank you, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Να επιχειρήσω να απαντήσω όσο μπορώ στις ερωτήσεις που έχουν τεθεί για τις κοινέ προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΠΕΣΚΟ. Ναι, είναι βασικό θέμα. Βέβαια, θα το δούμε του χρόνου που θα κάνουμε την ε, αναθεώρηση της ΠΕΣΚΟ. Όπως είπατε είναι λίγο νωρί. Είμαστε ακόμη σχετικά νέα πρωτοβουλία. Αλλά Ήδη έχουμε διαπιστώσει ορισμένα πρώτα θέματα όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων. Κάποια θετικά, μια θετική δυναμική από πλευρά πόρων από του εθνικού αμυντικού προπολογισμού, αλλά τα κράτη-μέλη καταλαβαίνουν ότι θέλει χρόνο για να έχουμε αποτελέσματα, για να αναπτύξουμε τι ε, δυνατότητε. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, στην εφαρμογή, το τελικό αποτέλεσμα. Και να το κάνουμε αυτό, τα κράτη-μέλη πρέπει να βάλουν αυτές τις ενωσιακές δυνατότητες στον εθνικό τους προγραμματισμό και αυτό από τη φύση του παίρνει χρόνο. Τα Υπουργεία Άμυνα, οι ένοπλε δυνάμει να βάλουν στον προγραμματισμό του πέρα από τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ και αυτή τη συμμετοχή τη ΠΕΣΚΟ. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα που το τονίζουμε στις συζητήσει. Για να βοηθήσουμε να έχει αυτά αποτελέσματα η ΠΕΣΚΟ. Για τη σχέση με το Ταμείο Άμυνα. Μα είναι βασικό θέμα για να υπάρχει μια ευρύτερη συνέπεια της εργασίας μας. Πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν διαφορετικές νομικές βάσεις βέβαια. Η ΠΕΣΚΟ είναι θέμα πολιτικής εξωτερικών και άμυνας, ενώ το Ταμείο Άμυνας είναι, βασίζεται στην ε, ενιαία αγορά. Η συνεργασία για τα προγράμματα της ΠΕΣΚΟ είναι μεταξύ των συμμετεχών των κρατών μελών, μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας, των Ενόπλων Δυνάμεων. Ενώ το Ταμείο Άμυνας βασίζεται σε επιχειρήσεις και βιομηχανικά, βιομηχανικούς ομίλους που ζητάνε χρηματοδότηση. Αλλά το βασικό είναι να εστιάζουμε στους ίδιους τομείς δυνατοτήτων. Οι προτεραιότητες ε, του οργανισμού άμυνας, της αρχής άμυνας, είναι το ζωτικό. Αλλά επειδή οι νομικές βάσεις είναι διαφορετικές, δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα ΠΕΣΚΟ για να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Άμυνα. Μπορεί να είναι διαφορετικέ αυτέ οι διαδικασίε. Αλλά Εάν θέλεις χρηματοδότηση από το Ταμείο για ένα πρόγραμμα που επίσης προωθείται από την ΠΕΣΚΟ, έχουμε ένα μπόνους 10% χρηματοδότηση επιπλέον. Υπό τον έλεγχο των συναδέλφων της Κομισιόν, βέβαια τα όλα αυτά που δεν είναι παρόντα σήμερα. Τώρα, όσον αφορά άλλους εταίρους για τα προγράμματά μας. Πολύ σημαντικό θέμα. Διεξάγεται τη συζήτηση για τα θέματα αυτά από τα κράτη-μέλη. Πρώτον, το κάθε μεμονωμένο πρόγραμμα θα έχει ή όχι εταίρους συνδεδεμένα κράτη-μέλη. Δεν έχει κανείς δικαίωμα να θεωρήσει ότι πρέπει να συμμετάσχει. Όχι, εμείς μπορεί να προσκαλέσουμε κάποιους να συμμετάσχουν. Τα προγράμματα επίσης βοηθάνε να εφαρμοστούν οι δεσμεύσει που έκαναν τα κράτη-μέλη, που ανέλαβαν συλλογικά η μεν εναντί των δε. Οπότε, η συμμετοχή και τρίτων χωρών σε αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να γίνεται αν υπάρχει συμπληρωματικότητα, αν δεν είναι προστιθεμένη αξία. Θα πρέπει να συμμερίζονται τις αξίες της Ένωσης. Υπάρχουν μια σειρά από νομικά κριτήρια, μια σειρά από προϋποθέσεις λοιπόν που τώρα τις καθορίζουμε. Τα κράτη-μέλη τις καθορίζουν και ελπίζουμε το Συμβούλιο να αποφασίσει στο εγγύς μέλλον επ' αυτών. Και όταν ληφθεί αυτή η απόφαση θα έχουμε λοιπόν και τις συνθήκες και τις διαδικασίες ούτως ώστε να ξεκινήσουν τα προγράμματα, να δούνε ποιοι εταίροι θα πληρώνουν αυτά τα κριτήρια, επί της ουσίας πολιτικά και νομικά. Άρα δεν έχει αποφασιστεί τίποτα, ελπίζουμε στο εγγύς μέλλον να γίνει κάτι τέτοιο, όταν θα ληφθεί η σχετική απόφαση, τότε τα μεμονωμένα προγράμματα θα δούνε. Θα καλέσουμε και συγκεκριμένους εταίρους τρίτες χώρες. Τώρα, πεδίο εφαρμογή των προγραμμάτων θα πούν και άλλοι συνάδελφοι. Πολλά είναι ανάπτυξη δυνατοτήτων, σχεδιασμός τεχνολογιών, νέοι εξοπλισμοί κτλ. Αλλά στο μέλλον θα έχουμε και λειτουργικά προγράμματα. Δηλαδή οι δυνατότητες που θα έχουμε θα πρέπει να συνδυάζονται, να έχουμε κοινή εκπαίδευση, κοινέ δομέ. Και θα γίνει όλο και πιο σημαντικό αυτός, αυτός ο τομέας. Αυτό θα βοηθήσει από την ίδια τη φύση του και την διαλειτουργικότητα. Οι συνάδελφοι θα πούν περισσότερα, υποθέτω. Η διαλειτουργικότητα βέβαια έχει πολλά επίπεδα. Είναι πολύ τεχνικό θέμα. Συνδεσιμότητα, για παράδειγμα, αλλά επίση ε, προδιαγραφέ και εκπαίδευση. Μία δέσμευση τη ΠΕΣΚΟ είναι η τυποποίηση. Και επίση να αξιοποιήσουμε και τι προδιαγραφέ του ΝΑΤΟ όσο γίνεται. Δεν θέλουμε δηλαδή να επανοπινεούμε τον τροχό κάθε φορά. 22 από τα 28 κράτη-μέλη είναι, όπως ξέρετε, και μέλη του ΝΑΤΟ και στα πλαίσια της ΠΕΣΚΟ είναι βέβαια 20 από τα 25. Άρα υπάρχει μια φυσιολογική εναρμόνιση με τον ΝΑΤΟ και τις προδιαγραφές του. Για την υποβολή εκθέσεων. Ε, είναι νωρίς ακόμη βέβαια. Αλλά νομίζω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων. Βέβαια, ακόμη μαθαίνουμε πώς να είναι πιο λεπτομερής η εκθέση μας. Είναι πολύ τεχνικής φύσης ε, να έχουμε όλα τα στοιχεία στη διάθεσή μας από τα εθνικά προγράμματα έρευνας. Αλλά νομίζω ότι τα πάμε καλά. Συγχρονισμός τώρα και συνεργασία των δομών άμυνας των διαφόρων κρατών μελών είναι πολύ περίπλοκο. Δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, θέλει χρόνο. Με τις δεσμεύσεις της ΠΕΣΚΟ και τα προγράμματα της ΠΕΣΚΟ τώρα έχουμε το μηχανισμό που θα επιτρέψει μία ευθυγράμμιση των διαδικασιών, κοινά εργαλεία λοιπόν για να εξολογούμε και την πρόοδο. Έχουμε λοιπόν ε, τα εργαλεία, τα μέσα, αλλά θέλουν χρόνο τα κράτη-μέλη για να τα εντάξουν όλα αυτά στον προγραμματισμό τους για να έχουμε αυτά αποτελέσματα, αλλά νομίζω πως και εδώ τα πάμε καλά. Τώρα για τα προγράμματα, δεν ξέρω αν σας έδωσα λάθος εντύπωση. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Κοιτάξτε, βέβαια ορισμένες φορές ε, κάποιοι είναι ανυπόμονοι. Αλλά τα πράγματα θέλουν το χρόνο τους. Για παράδειγμα, να δημιουργήσουμε μια κοινή υγειονομική δομή. Θέλει χρόνο για να σχεδιάσουμε νέους, ε, νέο εξοπλισμό για τα διάφορα προγράμματά μας. Αλλά η συνολική πρόοδος νομίζω είναι καλή. Αλλά και τα κράτη-μέλη τονίζουν ότι πρέπει να πιεστούμε περισσότερο για να εφαρμόσουμε τις δεσμεύσεις μας. τι συζήτηση έγινε στο Brussels 2. Είναι μια εκδήλωση την οποία δεν διοργανώσαμε εμείς, αλλά γενικά τα προγράμματα της ΠΕΣΚΟ λειτουργούν με βάση διάφορες ομάδες κρατών μελών και χρηματοδοτούνται από τις ομάδες κρατών μελών που συμμετέχουν. Άρα αυτοί αποφασίζουν τι θα χρηματοδοτήσουν ίσως αξιοποιώντας και χρηματοδότηση του Ταμείου Άμυνας ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω άλλων μηχανισμών. Τα προγράμματα λοιπόν τα τρέχουν, διάφορες ομάδες κρατών μελών υποβάλλουν εκθέσεις σε εμάς, αλλά την ευθύνη την έχουν αυτοί που τα τρέχουν. Το γενικότερο θέμα της στρατιωτικοποίησης κτλ. Δεν νομίζω ότι τώρα είναι η στιγμή να κάνουμε την πιο γενική αυτή συζήτηση, αλλά η ΠΕΣΚΟ είναι τμήμα της συνθήκης και έχει να κάνει με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Οποιαδήποτε χρήση στρατιωτικών δυνάμεων θα βασίζεται στις αρχές των συνθήκων. Πλήρη σεβασμό του Διεθνού δικαίου, για παράδειγμα. Τώρα, πόσο φιλόδοξοι είμαστε. Ναι, είναι θέμα συζήτηση, βέβαια. Αυτό πρέπει να την κάνουμε του χρόνου αυτή τη συζήτηση. Αλλά έχει καθοριστεί το επίπεδο φιλοδοξία από το Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2016 υπάρχουν προτεραιότητε, να ανταποκρινόμεθα σε σειράξει και κρίσει, να βοηθήσουμε του εταίρε μα να αναπτύξουν τι δικέ του δυνατότητε και τρίτον να προστατεύσουμε την Ένωση και του πολίτε τη. Αυτή είναι η βασική στόχη που έχει θέσει η ΠΕΣΚΟ. Για να έχουμε λοιπόν αυτό που αποκαλούμε ένα συνεκτικό πακέτο δυνάμεων, χωρί κενά, να έχουμε τι δυνατότητε που έχουμε για να εκτελέσουμε ορισμένε αποστολέ. Ένα δώσω τώρα το λόγο και του συναδέλφου ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά σημεία ήδη απαντήθηκαν και αναλυτικά. Δεν θα επαναλάβω όλα. Θα εστιαστώ επί των σημείων που αφορούν περισσότερο την υπηρεσία μας. Όσον αφορά τα κοινά προβλήματα, πράγματι αντιμετωπίζουμε πολλές νέες πρωτοβουλίες που θέτουν δύο προκλήσεις για τα κράτη-μέλη πρώτα απ' όλα να εξοικειωθούν με τους νέους μηχανισμούς και να επιβληθεί μια, μια συνοχή στους μηχανισμούς. Επιβάλλεται να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια τα κάτι μελη Εμείς, σαν φορέας, θέλουμε να βοηθήσουμε στο βαθμό του δυνατού τις χώρες όσον αφορά τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τον νέο μηχανισμό και με την αναγκαία συνοχή που όλοι επιδιώκουμε στους διάφορους ε, μηχανισμούς, στι διάφορες πρωτοβουλίε. Αυτό είναι ο κοινό στόχο η κοινή πρόκληση. Να φτάσουμε σε μια ταχύτητα πορεία, όπου οι μηχανισμοί να μην θεωρούνται σε κάτι εξωτικό, κάτι καινούριο, αλλά κάτι που υπησέρχεται στην πρακτική αναπτύξεως δυνατοτήτων των κρατών μελών στο σχεδιασμό του σε εθνικό επίπεδο, κάτι που θα γίνει φυσικό η χρήση αυτών των μηχανισμών και θα επιδιώξουν την συνοχή που είναι κοινό στόχο, χρησιμοποιώντας όλα τα εργολεία διευκόλυνση που του προσφέρονται και η Ευρωπαϊκή ε, Υπηρεσία Άμυνα αποτελεί ένα τμήμα αυτού. Πάω τώρα στο άλλο ερώτημα που αφορά τα 34 προγράμματα. Δίκιο έχετε. Κάποια από τα προγράμματα ε, τίνουν περισσότερο από την έρευνα και ανάπτυξη αλλά στατιωτική δυνατότητα τι εννοούμε. Εννοούμε ένα σύνολο μέσων που αναπτύσσονται και εντάσσονται σε ένα περιβάλλον που επιτρέπει τη χρήση τους. Στο ΝΑΤΟ χρησιμοποιούμε μια λέξη κάπως δύσκολη OTM, NPF, ε, δηλαδή αποτελείται από το δόγμα χρήσεως του υλικού εκπαίδευση όσον αφορά ε, τη διαδικασία και το λογισμικό για τη χρήση του εξοπλισμού. Κανένα πεδίο δεν είναι κλειστό όσον αφορά τη μόνιμη συνεργασία, τη διαθρωμένη. Και έχουμε διαδικασίες που καλύπτει αυτού του τομεί σήμερα, που καλύπτουν προγράμματα που αφορούν την κοινή οργάνωση όσον αφορά τη χρήση συγκεκριμένων δυνατοτήτων. Έχουν προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση έχουν προγράμματα που αφορούν λίγο τη διλειτουργικότητα, ακόμα και αν δεν υπάρχουν πολλά τέτοια προγράμματα και έχουν προγράμματα που όλο και περισσότερο αφορούν το υλικό. Είναι, ε, η ΠΕΣΚΟ είναι καινούργια πρωτοβουλία. Τα κάτι μελη χρησιμοποίησαν τις δύο πρώτες ομάδες προγραμμάτων για να υλοποιήσει το μηχανισμό και δημιουργείται μια κάποια οριμότητα και είμαι σίγουρος ότι όλο και περισσότερο θα έχουμε προγράμματα τα οποία θα είναι πιο καλά στοχευμένα σε αυτά τα προγράμματα υπάρχει ένα διακύβευμα. Ο συγχρονισμός με τα προγράμματα τα εθνικά αναπτύξεως δυνατοτήτων. Και εκεί το CARD είναι σημαντικό μέσο, είναι στα χέρια των κρατών μελών για να μπορέσουν να εντάξουν στον εθνικό του σχεδιασμό στόχους συνεργασίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί ο συγχρονισμός μεταξύ ΠΕΣΚΟ και CARD είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ξεκινάμε τον πρώτο πλήρη κύκλο του CARD αυτή τη στιγμή. Ο οργανισμός επισκέπτεται τα κράτη-μέλη για να προβεί σε διάλογο με θέμα το μηχανισμό CARD. Και αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει βέβαια να βοηθήσει τα κράτη-μέλη ούτως ώστε τελικά τα κράτη-μέλη να θέσουν στόχους όσον αφορά την ανάπτυξη δυνατοτήτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενταχθούν αυτοί οι στόχοι στον εθνικό σχεδιασμό και αυτοί οι επιλεγέντες στόχοι που θα ενταχθούν θα οδηγήσουν σε υποβολή προτάσεων για προγράμματα ΠΕΣΚΟ. Συγχρονισμός και συνοχή είναι κάτι που ζητούμε και επιδιώκουμε. Ο πρώτος κύκλος του ΚΑΡΔ ξεκινά και θα δώσει τη δυνατότητα στα κάτι μελη να εξοικειωθούν με αυτή τη διαδικασία ούτως ώστε να καταλήξουμε στον αναγκαίο ε, συγχρονισμό και στη συνοχή. Πάνω σε αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικός απολογισμός. Αυτό προσπάθησα να πω στην αρχική μου παρέμβαση. Δεν έχουμε μόνο μικρά προγράμματα. Έχουμε κάποια προγράμματα ήδη τα οποία είναι αρκετά σημαντικά και μεγάλα. Δεν θα τα σχολιάσω εγώ. Ο οργανισμός μας υποστηρίζει τα κράτη-μέλη και δεν σχολιάζουμε τα προγράμματα των κρατών μελών και θα με εξέπλητε αν δεν έβρισκα πιο μεγάλα προγράμματα να προτείνονται στο μέλλον. Όσον αφορά τις φιλοδοξίε των κρατών μελών και τις φιλοδοξίε τη ΠΕΣΚΟ, εξαρτάται από τι επίπεδο φιλοδοξιών έχουν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν στα πλαίσια του μονίου μηχανισμού. Πάντως έχουμε μπει στη... είναι καλή η πορεία που ακολουθούμε και τα πράγματα πάνε σε μια τάξη. Ευχαριστώ. Ο λόγος του κύριου ε, with my turn. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένα από τα ερωτήματα. Για το πρώτο, πώς η εφαρμογή της ΠΕΣΚΟ μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική. Ως γραμματεία ΠΕΣΚΟ έχουμε διεξάγει διμερείς συναντήσεις με τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν και μετά από δικό τους αίτημα τις αρχές Ιουνίου μέχρι τον Οκτώβριο έχουμε κάνει συναντήσεις με τα κράτη-μέλη σε διμερές επίπεδο. Συζητήθηκαν διάφορα, ανάμεσα στα οποία και το πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή των εθνικών σχεδίων. Ποιους τρόπους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εφαρμοστεί τελικά η ΠΕΣΚΟ έκαναν κάποιε προτάσει στα κράτη-μέλη, τις οποίες λαμβάνουμε υπόψη μα για την στρατηγική που θα καταρτήσουμε για τον επόμενο χρόνο. Έχει ήδη απαντηθεί η σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και η σχέση μας με τρίτες χώρες. Θα σταθώ λίγο περισσότερο στο θέμα της διαλειτουργικότητας. Στην πρωτολογία μου ανέφερα ότι η διαλειτουργικότητα είναι μία από τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί και την εξετάζουμε ενδελεχώς από πλευρά στρατιωτικής. Οποτεδήποτε μας υποβάλλεται μια πρόταση για ένα έργο, εξετάζουμε και δίνουμε μεγάλη προσοχή στο κατά πόσο μπορεί αυτό το έργο να συνεισφέρει στη διαλειτουργικότητα είναι πολύ σημαντικό για να επιτύχει κανείς την αποστολή του, να επιτύχουν οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ευρώπης την αποστολή τους, να μπορούν να ακολουθούν τα ίδια δόγματα, να έχουν αντίστοιχη εκπαίδευση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν επιδιώκουμε την τυποποίηση και γενικότερη διαλειτουργικότητα υπό το γενικό τίτλο της δέσμευσης 13 που έχει τον τίτλο διαλειτουργικότητα. Υπάρχουν και συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία αναφέρονται ιδιαίτερα στο θέμα της εκπαίδευσης των στελεχών που εκ πρώτης όψεως μπορεί να μην αντιλαμβάνεται κανείς πώς συνεισφέρουν στη διαθεσιμότητα και τη διαλειτουργικότητα όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο, πραγματικά συνεισφέρουν στη διαλειτουργικότητα. Τη λαμβάνουμε λοιπόν υπόψη μας πάρα πολύ ε, σοβαρά την διαλειτουργικότητα. Θεωρούμε κρίσιμη σημασία. σε σχέση με προγράμματα ΠΕΣΚΟ τα οποία ολοκληρώθηκαν ή σταμάτησαν. Εξ όσων γνωρίζω δεν έχει ακυρωθεί, δεν έχει διακοπεί κάποιο project ΠΕΣΚΟ. Έτσι κι αλλιώς είναι στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά από όσο γνωρίζω και η πρώτη δέσμη και η δεύτερη δέσμη έργων συνεχίζεται να υλοποιείται. Μέχρι το 2022 περιμένουμε να έχουν υπάρξει δηλώσεις για τις επιχειρησιακές δυνατότητες από 12 από αυτά τα project. Αυτά από την πλευρά μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Λίγη συνεδρίαση μας. Okay. Good morning. Ωραία, καλημέρα σας αγαπητοί συναδελφοί. Να συνεχίσουμε γιατί έχουμε καθυστέρηση. Σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Στρατιωτική κινητικότητα. Πώς έχουν τα πράγματα και ποιες είναι οι προοπτικές. Να καλωσορίσει και πάλι στους συγκεκριμένους μας τον κύριο Φρανκ Ντεζίτε και τον κύριο Αρνού Μόλενάρα που τους έχουμε ήδη από προηγουμένως και να σας δώσω το χρόνο να καθίσετε ο κύριος Ζωαλουί Κόλσον που είναι επικεφαλής της ε, μονάδας για τα δίκτυα μεταφορών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχει στην εργασία για τη στρατηγική κινητικότητα που είναι τμήμα του προγράμματος Συνδέοντας την Ευρώπη και ασχολείται με τι απαιτήσει τη διπτής χρήση. Η βελτιότητα τη στρατηγικής κινητικότητας είναι βασική πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμβάλλει στην ε, εφαρμογή των φιλοδοξιών μα στον τομέα τη ασφάλεια και άμυνας όπω την, κατά, την στο ε, Συμβούλιο. Σήμερα η Επιτροπή μας ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις πρόσφατες εξελίξεις για το θέμα αυτό και πολύ συγκεκριμένα θέματα όπως η μεταφορά επικίνδυνων ουσιών ή ο συντονισμό με τον ΝΑΤΟ. Γι' αυτό σας παρακαλώ εξηγήστε μας πώς πάνε τα προγράμματά σας, Ποιε δράσεις θα πρέπει να υιοθετηθούν στο μέλλον. Λοιπόν, θα έλεγα να πάρει πρώτα το λόγο ο κύριος Κολσούν, μετά ο κύριος Ντεζίτ και μετά ο κύριος Μόλεναρ. Κάθε παρέμβαση παρακαλώ 10 λεπτά για να έχουμε χρόνο και για έρωτα απαντήσεις. Προβλέπετε το θέμα αυτό μέχρι τις 11 η ώρα. Εάν υπάρξει κάποια μικρή υπέρβαση, ε, καλώς. Αλλά σας παρακαλώ να τηρείτε το δεκάλεπτό σας. Ο κύριος Χολσόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που οργανώσατε αυτή τη συζήτηση για ένα θέμα που είναι σίγουρα σημαντικό. Είναι πρωτοβουλία της πολιτικής άμυνας θεμελιώδου σημασίας και για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα είμαι πολύ σύντομος να επενθυμίσω το πλαίσιο αυτού του προγράμματος δράσης. Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος Ιούνκερ είπε πόση σημασία έχει η δημιουργία της Ευρώπης της άμυνας. Στα πλαίσια αυτά, βεβαίως, παίζει μεγάλο ρόλο η στρατιωτική κινητικότητα. Κινητικότητα των στρατιωτικών. Τα τελευταία χρόνια έχουμε εφαρμόσει τις τέσσερις ελευθερίες, ε, την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, των κεφαλαίων κτλ. Αλλά η ίδια στρατιωτική δεν μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στα πλαίσια της Ένωσης. Είναι μια πρόκληση λοιπόν. Από δύο απόψεις. Από τη μία, διότι αν υπάρξει μια εξωτερική απειλή, η ελεύθερη κυκλοφορία των ενόπλων δυνάμεων δεν μπορεί να γίνει εύκολα και επαρκώς. Και από την άλλη πλευρά, όταν θέλουμε να στείλουμε δυνάμεις εκτός της Ένωσης για κάποιες επιχειρήσεις που τις γνωρίζετε και εδώ έχουμε προκλήσεις ούτω ώστε οι δυνάμεις μας να μπορέσουν να αποσταλούν εκεί που χρειάζονται. Έχουμε λοιπόν αυτές τις προκλήσεις. Η Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης εντόπισαν δύο ειδών εμπόδια. Ορισμένα είναι νομικής και κανονιστικής φύσης. Για παράδειγμα, χρειάζονται εγκρίσεις, ούτω ώστε στρατιωτικοί να πάνε από το ένα σημείο στο άλλο. Υπάρχουν διαφορετικές νομοθεσίες. Για παράδειγμα, για τις επικίνδυνες ουσίες. Όταν στρατιωτικές αυτοκινητοπομπές περνάνε σύνορα, υφίστανται διαφορετικοί κανόνες. Υπάρχουν τελωνιακά θέματα, δεν έχουν ρυθμιστεί φορολογικά δεν έχουν ρυθμιστεί. Όλα αυτά αποτελούν ουσιώδη εμπόδια για να μπορεί να υπάρχει αυτή η κινητικότητα. Και ο δεύτερος τομέας είναι τα φυσικά εμπόδια. Οι δομές δεν είναι πάντα προσαρμοσμένες. Οι υποδομές. Και η γνώση των ε, στοιχείων των υποδομών επίσης δεν είναι πάντα γνωστή. Δεν, πάντα, δεν υπάρχει πάντα. Το πρόγραμμα δράσης της 28ης Μαΐου 2018 προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματα αυτά. Εσκεμένα εστιάζει σε ένα περιορισμένο αριθμό δράσεων για να αντιμετωπίσει ή να μειώσει τα προβλήματα που ανέφερα και δεύτερο χαρακτηριστικό του εστιάζει επιδράσεων όπου υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες με τις ευρωπαϊκές κοινέ πολιτικές. Θέλουμε να βασιστούμε στις ευρωπαϊκές κοινέ πολιτικές στο μη στρατιωτικό τομέα για να δημιουργήσουμε, να ευνοήσουμε αυτήν την κινητικότητα των στρατιωτικών ή του στρατιωτικού τομέα γενικότερα. Τώρα, όσον αφορά τις υποδομές με τις οποίες θα ασχοληθώ, είχαμε καθορισμό ενιαίων προδιαγραφών για τις στρατιωτικές υποδομές ενεκρίθησαν σε επίπεδο Ένωσης και επίσης το ίδιο έγγραφο καθορίζει και τα δρομολόγια που θα πρέπει να ακολουθούν για τα στρατιωτικά οχήματα στην κυκλοφορία τους. Σε αυτή τη βάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έκανε μια πρώτη δουλειά, δηλαδή να εξετάσουν τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των στρατιωτικών υποδομών που ενεκρίθησαν από τη μία και από την άλλη τις ε, πολιτικές υποδομές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Να δουν ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Και επίσης, ποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ των στρατιωτικών χαρτών που έχουν εγκριθεί και των χαρτών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Και έχουμε ήδη κάποια αποτελέσματα. Τα Ναι, μεν υπάρχουν διαφορές. Αλλά δεν είναι τόσο σημαντικές όσο θα μπορούσε να υποθέσει κανείς. Και για τους χάρτες. κατά 94% συμπίπτουν με τους χάρτες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Άρα μπορεί να υπάρχει συνδυασμός μεταξύ των πολιτικών και αμυντικών πολιτικών στον τομέα που μας ενδιαφέρει. Τρίτον, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπεριέλαβαν στο μηχανισμό διασύνδεσης της Ευρώπης που χρηματοδοτεί τις υποδομές μεταφορών συμπεριέλαβαν λοιπόν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν υποδομές μεταφορών διτής χρήσης. Τι σημαίνει αυτό. Υποδομές μεταφορών που θα κατασκευαστούν για τις στρατιωτικές ανάγκες αλλά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και για τις πολιτικές μεταφορές. Υπήρξε συμφωνία Κοινοβουλίου Συμβουλίου στις 7 Μαρτίου 18 επ' αυτού. Θα υπάρχει δυνατότητα μέσω του μηχανισμού συνδέοντας την Ευρώπη να χρηματοδοτηθούν υποδομές μεταφορών να κατασκευαστούν ή να βελτιωθούν κάποιες υποδομές για στρατιωτική χρήση που να έχουν επίσης χρησιμότητα για, την, ε, για τις πολιτικές μεταφορές. Αυτή είναι η δυτή χρήση. Θέλουμε τώρα να καθορίσουμε πού θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοιες υποδομές δυτής χρήσης. Συζητάμε τα κράτη-μέλη. Έγινε μια πρώτη συνάντηση στις 27 Σεπτεμβρίου. Θα γίνουν δύο ακόμη, μία το Δεκέμβριο και η επόμενη τον Ιανουάριο. Και θεωρούμε ότι μετά από αυτές τις τρεις συνεδριάσεις θα καταλήξουμε σε συμφωνία με τα κράτη-μέλη επί των ορισμών στον τομέα αυτό της χρήσης. Δηλαδή, μέχρι ποιο επίπεδο μπορούμε να χρηματοδοτούμε υποδομές μεταφορών για να είναι χρήσιμες για τις στρατιωτικές μεταφορές, αλλά να έχουν και μία χρησιμότητα για τις πολιτικές μεταφορές. Η επόμενη φύση θα έχει να κάνει με το πολιετές δημοσιονομικό 2127, όπου το Κοινοβούλιο σίγουρα θα παίξει πλήρως το ρόλο του. Η Επιτροπή πρότεινε ένα προϋπολογισμό 6,5 δις για την στρατιωτική λοιπόν κινητικότητα και ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί αυτό το κονδύλι, ότι θα συμφωνήσουν Κοινοβούλιο-Συμβούλιο από αυτού στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαίσιου. Κατά λίγο. Για τις υποδομές. Με το εξής. Αυτή η πρωτοβουλία για την στρατιωτική κινητικότητα είναι πολύ σημαντική για τις υποδομές μεταφορών γιατί είναι μια πρωτοβουλία όπου όλοι κερδίζουμε. Θα χρηματοδοτήσουμε και θα κατασκευάσουμε υποδομές που είναι αναγκαίες για τις στρατιωτικές μετακινήσεις. Άρα κάνουμε κάτι, χρήσουμε, ε, θα κάνουμε κάτι χρήσιμο για τον ε, πυλώνα το στρατιωτικό, αλλά θα έχουν τι χρήση οι υποδομές αυτές. Θα βοηθήσουμε λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών να ολοκληρωθεί πιο σύντομα. Θα βοηθήσουμε το δίκτυο αυτό να ολοκληρωθεί πιο σύντομα. Άρα κερδίζουν όλοι. Πολλές ευρωπαϊκές πολιτικές. Γιατί συμβάλλουμε παράλληλα και στην πολιτική άμυνα και στην πολιτική μεταφορά. Υπάρχουν και άλλοι δομείς στο πρόγραμμα δράσης για παράδειγμα τελωνιακά θέματα, επί των οποίων ε, η Επιτροπή έχει σημειώσει ουσιώδη πρόοδο και φορολογικά, όπου προβλέπεται ιδιαίτερα ο ΦΠΑ. Οι στρατιωτικές ασκήσεις στα πλαίσια του ΝΑΤΟ εξαιρούνται από το ΦΠΑ και θέλουμε να το διευρύνουμε αυτό στις στρατιωτικές ασκήσεις που γίνονται στα πλαίσια της κοινή πολιτικής άμυνας. Έγινε μια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Συμβούλιο για το θέμα αυτό τον περασμένο Μάρτιο και ελπίζουμε να την εγκρίνει το Συμβούλιο όσο ταχύτερα γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Κωσό. Έχετε το λόγο κύριε Δεσίβ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να σας θα συμπληρώσω αυτή την παρουσίαση και θα εστιαστώ επί του πρόοδου που έχουμε πετύχει ε, στα πλαίσια τη υπηρεσία εξωτερική δράση και την κινητικότητα, κατά πόσο ταιριάζει και στο σχέδιο δράση που παρουσιάστηκε στι 28 Μαρτίου του Μαρτίου του 2018 για τη θετική κινητικότητα. Θέλουμε αποτελεσματική και έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά στατιωτικού προσωπικού και των διαφόρων μέσων για να καλυφθούν οι ανάγκε τη Ευρωπαϊκή Ενώση στα πλαίσια επιχειρήσεων και ασκήσεων και για οποιαδήποτε καθημερινή μετακίνηση. Καλύτερη κινητικότητα των δυνάμεων εντό και πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια, διότι τα κράτη-μέλη θα μπορούν να δράσουν ταχύτερα σύμφωνα με τι διάφορε ανάγκε και ευθύνε που έχουν, πολύ συχνά στα πλαίσια αποστολών και και επιχειρήσεων, καθώ και επίπεδο εθνικό και πολυεθνικό. Η στρατιωτική κινητικότητα καλύπτει τη μετακίνηση στρατιωτικού προσωπικού και μέσων από μία τοποθεσία σε άλλη, συμπεριλαμβανομένη και τη διέλευση συνόρων, η χρήση διαφόρων τρόπων μεταφορά. Η στρατιωτική κινητικότητα αυτή καθεαυτή δεν είναι μια δυνατότητα, αλλά είναι κάτι που ε, διευκολύνει τι δραστηριότητε. Αυτή η κινητικότητα, η στατιωτική, είναι εθνική ευθύνη. Ο σχεδιασμό και η εκτέλεση συμπεριλαμβάνεται σε αυτό και έγκαιρη παροχή εξοπλισμού, υπηρεσιών και υποδομών. Λόγω της αποκλειστικού, του αποκλειστικού πολυεθνικού χαρακτήρα των, υπηρεσιών, των επιχειρήσεων ΚΕΠΑ, χρειάζεται συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. Η στατιωτική κινητικότητα έγινε θέμα που υψηλού πολιτικού ενδιαφέροντος του 2016, Διότι τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω κατάλαβαν τότε τι δυσκολίε που αντιμετωπίζονται τη μετακίνηση στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη κατά διάρκεια περίοδου ειρήνη. Και γι' αυτό δημιουργήσαμε μια ομάδα εργασία για να εντοπίσουμε τι δυσκολίε που υπάρχουν όσον αφορά αυτό το θέμα και να λάβουμε υπόψη διάφορε εμπειρίε των εξωτερικών φορέων όπω είναι το ΝΑΤΟ, η ΙΠΑ ή ο Καναδά. Έτσι, το 2017 και το 2018 Δημιουργήσαμε έναν οδικό χάρτη για διασυνοριακή μεταφορά στρατευμάτων. Το σχέδιο δράση Ευρωπαϊκή Ενώσεω βασίζεται στον οδικό χάρτη αυτό και παρέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε τα εντοπιστέτα προβλήματα σε συντονισμένο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι βασικέ δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση που καθορίζουν το σχέδιο δράση που αφορούν τι θετικέ απαιτήσει για υποδομέ και μεταφορέ, ρυθμιστικά, κανονιστικά θέματα, διαδικαστικά, ε, ε, ΦΠΑ, ε, δασμούς και άδειες διελεύσεως συνόρων. Στα πλαίσια του δικού μας χάρτη, τα κράτη-μέλη ανέθεσαν στον οργανισμό να ε, θεσπίσει δύο προγράμματα πλαίσια. Το ένα για τη βελτιστοποίηση διασυνοριτικών αδειών για μετακινήσεις και διαδικασίες για αυτό το θέμα στην Ευρώπη και δεύτερον εναρμόνιση των στετικών ε, αναγκών όσον αφορά τα τελωνία. Επίση, ο οργανισμός θα έπρεπε να κάνει δύο ερευνές για επικίνδυνα ε, αγαθά και νομικές στοιχεία. Τα κράτη-μέλη ζήτησαν η EDA να συνεχίσει να παρέχει μια πλατφόρμα για ανταλλαγή απόψεων και η έκθεση προόδου ετησίω που θα υποβάλλεται ετησίω. Η πρώτη έκθεση ήδη υπευλήθη τον Μάιο νεστότο έτου στο Διοικητικό Συμβούλιο και συμβάλλει αυτές οι εκθέσεις ε, η έκθεση αυτή και στην έκθεση τσίπα τη εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να υπάρχει συμπληρωματικότητα όσον αφορά τι εκθέσει, κάτι προβλέπεται στο σχέδιο δράση. Αν επιτρέπετε, θα σα δώσω λεπτομέρειε δραστηριότητε αυτέ που ανέφερε. Το πρόγραμμα βελτιστοποίηση των διαδικασιών αδειοδότηση διαλέξεων συνόρων δημιουργήθηκε για να προωθηθεί η εναρμόνιση και απλούστευση διασυνοριακών μετακινήσεων σχετικών διαδικασιών, αντιμετωπίζοντας διαδικαστικά και ρυθμιστικά θέματα και προβλήματα, συνδυασμό με τις διάφορες διαδικασίες για αδειοδότηση, ελήψη εναρμονισμένη διαδικασίας μεταξύ κρατών μελών, διότι αυτή η εναρμόνιση, η έλλειψη εναρμόνιση εμπόδισε μεταφορά συνδευμάτων στην Ευρώπη. Ε, χερσαίες μεταφορές καλύψαμε, ενέργειες μεταφορές, ε, μεταφορά ε, των δυνατοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσει για διάφορες επιχειρήσεις. Τεχνικές διευθετήσεις για τη συνοριακή διέλευση από ξηρά και αέρα έχει σαν στόχο να βρούμε ε, κάποιους τομείς που πρέπει να γίνει εναρμόνιση σε αυτές τις μεταφορές. Οι διευθετήσεις έχουν υπογραφεί από 22 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής το 22 Μαρτίου του 2019 Πέραν αυτών τα κράτη-μέλη ξέρουμε ότι έχουμε 25 κράτη-μέλη που συμμετέχουν τώρα σε αυτή τη φάση. Ένα δεύτερο πρόγραμμα για τα τελωνία και τους δασμούς ε, καλύπτει διάφορες τελωνιακές δραστηριότητε και το πρόγραμμα αυτό έχει προχωρήσει σημαντικά. Όπως τα γνωρίζετε μέχρι τώρα, τα κράτη-μέλη βασιζόταν σε τελωνιακό έντυπο, το 402 του ΝΑΤΟ, για τη μεταφορά αγαθών ε, η χρήση αγαθών σε θετικέ επιχειρήσει, διότι δεν υπήρχε έντυπο αντίστοιχο στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Έτσι, δε περαιτέρω, ένα από τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με τα κράτη-μέλη και τρίτα μέρη ήταν ότι κάποιε δυσκολίε που αντιμετωπιστήκαν από του στρατιωτικού στη διέλευση των συνόρων απέρευσαν από την έλλειψη σαφήνεια ή απουσία κάποιων στοιχείων στο έντυπο του ΝΑΤΟ που χρονολογείται από τη δεκαετία του 50. Η στρατηγική κινητικότητα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω θέλουν να διευκολύνουν την ανάπτυξη δυνάμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πέραν τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για να υποστηριχθούν επιχειρήσει ΚΕΠΑ. Γι' αυτό τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να αναπτυχθεί ένα έντυπο τελωνιακό για στρατηγικού σκοπού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που αναφέρεται στο σχέδιο δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε λιγότερο από έξι μήνες, οι στατιωτικέ αρχές συνέκλειναν σε μια τυποποιημένη διαδικασία για τελωνιακέ διαδικασίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δημιουργία ενός εντύπου μιας μορφής, ενός μορφοτύπου κοινού. Και ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεση. Αυτή η προσπάθεια δεν εμποδίζει να χρησιμοποιήσουμε την, ε, το έντυπο του ΝΑΤΟ. Από πλευρά νομική το έντυπο του ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή, το έντυπο τη Ευρωπαϊκή Ενώσης θα είναι ξεχωριστά. Θέλουμε να ευθυγραμμίσουμε του μορφότυπου Ευρωπαϊκή Ενώσης και του ΝΑΤΟ και να χρησιμοποιούμε ταυτόσημα έντυπα. Ε, δε, ο συντονισμός προσωπικού δεν οδήγησε σε θεώρηση πλευρά του ΝΑΤΟ, αλλά ελπίζουμε ότι θα φεγραμιστεί το έντυπο του ΝΑΤΟ, λαμβάνοντας ε, την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται από την αναθεώρηση για τι ανώπιε έχει ψηφιοποιηθεί το έντυπο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως, κάτι που συμπονήθηκε από του αρμόδιου φορεί τον Αύγουστο. Και το είπε και ο συνάδελφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τεθεί σε ισχύ αυτό το έντυπο όταν η αναθωρημένο τελωνιακός κώδικα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως θα δημοσιευτεί. Άλλε προσπάθειε που γίνονται στο πρόγραμμα σχετικά με τελωνιακά αφορούν την ψηφιοποίηση των τελωνιακών διαδικασιών μέσω τη υιοθέτηση τελωνιακού κώδικα Ευρωπαϊκή Ενώσεω του Μαίου του 2016, που αντικαθιστά τον κοινοτικό τελωνιακό κώδικα του 1992. Η ψηφιοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών ξεπερνά 2 εκατομμύρια ανταλλαγής εντύπων, φυσικών εντύπων και αυτό θα μειώσει και το χρόνο που θα πετύχει την ε, ολοκλήρωση τελωνιακών διατυπώσεων και του ελληνικού ελέγχου, και έτσι θα βελτιώσει τη στρατηγική κινητικότητα όλη αυτή η ψηφιοποίηση. Βάσει των παραμέτρων που ανέφερα, ο συντονισμό μεταξύ του φορέα μα και των κρατών μελών θα οδηγήσει σε εναρμόνιση των τελωνιακών διαδικασιών και για την ώρα μα σε αρχική φάση. Έχουμε αυτά τα δύο προγράμματα. Κάναμε δύο εκθέσει για τα επικίνδυνα αγαθά και τι νομικέ πτυχέ. Εξετάσαμε τι νομικέ πτυχέ που αφορούν σε εθνική κινητικότητα και είναι μια βασική δράση που απορρέει από εκεί και απορρέει από το σχέδιο δράση τη Ευρωπαϊκή Ενώση για τη εθνική κινητικότητα. Αυτή η έκθεση αναφέρεται στο εθνικό νομικό πλαίσιο για όλων των κρατών μελών και αποκλήσεις που υπάρχουν για το διεθνές και το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσης και Διδράσης ενετόπισε και το τι γίνεται με τους κανόνες που ισχύουν για τη μεταφορά επικινδύνων αγαθών στο θετικό τομέα και αυτό είναι ένας άλλος τομέας δράσης. Τα τελικά αποτελέσματα και συμπεράσματα των δύο ερευνών τα έχουν αποσταλεί στις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναφέρονται στην ετήσια έκθεση του 2019 περί στατιωτικής κινητικότητας. Να τονίσω ότι η Γενική Διεύθυνση MOVE τόνισε στο, στο διευθυντικό προσωπικό του CDA ότι η έκθεση συμπεραβάνει πολλές πληροφορίες που θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση ανάγκης για περαιτέρω δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει αυτή την εξέταση και την ανάλυση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περαιτέρω δραστηριότητε που απορρέουν από τι έρευνε αυτέ θα λάβουν χώρα στα πλαίσια των προγραμμάτων για διοδότηση διασυνοριακή διέλευση θετικών δυνάμεων. Θέλουμε να βελτιώσουμε η θετική κινητικότητα και το πρόβλημα να ιδωθεί με άλλε δραστηριότητε που έχουν δρομολογηθεί. Κάνουμε, ε, υλοποιούμε δύο προγράμματα για πολυτροπικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για διπλωματικές άδειες. Για τον πολυτροπικές μεταφορές έχουμε, βρει, έχουμε ένα πλαίσιο το 2013 και έχουμε θέσει ένα γεωγραφικό πλαίσιο μετακίνηση στατευμάτων. 14 κράτη-μέλη συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τεχνικέ διευθυντήσεις για τη διέλευση των συνόρων και τη μεταφορά χερσαίων ε, δυνάμεων. Είμαστε στο στάδιο υπογραφή. Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά προέγκριση για διπλωματική αδειοδότηση ε, εναερίων μεταφορών. Το 2012 ξεκίνησε η ανάλυση αυτή και τα 20 κράτη-μέλη έχουν υπογράψει τεχνικέ διευθυντήσει. Τα δύο προγράμματα χρησιμοποιούνται σαν βάση για δραστηριότητε εντό του προγράμματο διασυνοριακών μετακινήσεων και σχετικών αδειών. Εν γέννη, αντικατοπτρίζονται σε αυτέ οι διαδικασίε. Αν δούμε όλε τι διαδικασίε, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε επιτύχει ουσιαστική πρόοδο. Στο μέλλον, η σχετική κινητικότητα παραμένει η μακροπρόθεσμη προσπάθεια που απαιτεί Συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και συνεργασία αυτών. Οι δραστηριότητε τη CDA θα συνεχίσουν να ωφελούνται από τη δραστηριότητα των κρατών μελών, καθώ και στενή συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων. Σε συνοχή με τι πρωτοβουλίε του ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ. Εσύ. ευχαριστούμε κύριε Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και μια και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εγώ απλώ θα συμπληρώσω, θα προσθέσω κάποια στοιχεία. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι ε, έχει υπάρξει μια καλή, ε, καλό επίπεδο συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και του στρατιωτικού προσωπικού και των γενικών διευθύνσεων τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίω τη Γενική Διευθύνσης MOVE. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα στοιχείο που έχει συνεισφέρει στην πρόοδο που είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Το σχέδιο δράσης που ήδη αναφέρθηκε είναι αυτό που καθορίζει τις δράσεις που αναλαμβάνουμε στους διάφορους τομείς και που εξασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνεκτικότητα των ενεργειών μας. Τα προβλήματα που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε έχουν προκύψει από την εμπειρία που έχουν μοιραστεί μαζί μας τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουμε δηλαδή προβλήματα και περιορισμούς που έχουν ε, παρατηρηθεί στην ε, μετακίνηση των δυνάμεων, στην αύξηση του κόστου της μετακίνησης αυτής ή καθυστερήσεις. Λαμβάνουμε υπόψη μας βεβαίως τα εξής στοιχεία. Πρώτα απ' όλα ε, σεβόμαστε πλήρως την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών. Κάθε κράτος μέλος έχει απόλυτο έλεγχο ε, σε περίπτωση που υπάρχει μετακίνηση στρατιωτικών δυνάμεων ή εξοπλισμού μέσω του εδάφους του. Δεύτερο, προσπαθούμε να έχουμε μια συντονισμένη ε, προσέγγιση ε, μεταξύ της στρατιωτικής και, και, και του πολιτικού σκέλους. Τρίτο. Μια και έχουμε πολλέ δραστηριότητε, πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει συντονισμό και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο κρατών μελών. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Τέταρτη αρχή είναι η συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Ήδη αναφέρθηκε, γι' αυτό δεν θα επεκταθώ. Σε γενικέ γραμμέ θα έλεγα ότι τηρούμε και υλοποιούμε ε, επιτυχώ το σχέδιο δράση. Ε, το βλέπετε αυτό και στην έκθεση που υπέβαλε η υπατή εκπρόσωπο στο Συμβούλιο τον Ιούνιο. Η βάση για την κατάρτιση του σχεδίου δράσης είναι οι στρατιωτικές ανάγκες, ε, στις οποίες, οι οποίες συμφωνήθηκαν στη Στρατιωτική Επιτροπή του Συμβουλίου. Και όπως εξήγησε, και εξήγησε ήδη ο συνάδελφος από την Επιτροπή πώς έγινε αυτό, ότι έγινε μια ε, διαδικασία με την οποία εντοπίστηκαν τα κενά και τι πρέπει να γίνει για να τα καλύψουμε. Μετά ε, δόθηκαν κάποιες διευκρινήσεις ε, για τις στρατιωτικές ανάγκες και τον Ιούλιο έδωσε την τελική του έγκριση το Συμβούλιο. Υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες και ιδίω στον τομέα των, ε, του κανονιστικού πλησίου, της διασυνοριακής μετακίνησης επικίνδυνων αγαθών κτλ συμπληρωματικά προς τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί να διευκολύνουν αυτές τις μετακινήσεις στο δικό τους επίπεδο. Θα σας υπενθυμίσω ότι μία από τις δεσμεύσεις της ΠΕΣΚΟ αναφέρεται ακριβώς στη στρατιωτική κινητικότητα και υπάρχει υπάρξει και σχετικό έργο του οποίου συντονιστής είναι οι κατοχώρες. Και εκείνες θα παρουσιάσουν την ε, πρόοδο που είχε σημειωθεί, αλλά αυτό που κυρίως γίνεται μέσω αυτού του project PESCO ε, είναι να βλέπουμε τι πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο. Αναφέρθηκε και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου τα σχετικά πέρυσι. Λέγεται ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν εθνικά σχέδια δράσης, να επιτρέπουν την διέλευση την διασυνοριακή μέσα σε πέντε εργάσιμες μέρες, να δημιουργήσουν ένα, ένα δίκτυο εθνικών σημείων επαφής και επίσης να κάνουν και ασκήσεις ανταποκρίσεις σε κρίση. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια συμπληρωματικότητα ανάμεσα στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Η συνεργασία με το ΝΑΤΟ είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Αναφέρεται και στην κοινή ε, διακήρυξη, ε, ε, προέρχεται μάλλον και από την κοινή διακήρυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ έχουμε δημιουργήσει έναν διαρθρωμένο διάλογο για τη στρατιωτική κινητικότητα, στον οποίο συμμετέχει στρατιωτικό προσωπικό και από τη δική μας την πλευρά και από την πλευρά του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, εχθές έγινε μια συνάντηση αυτής της Επιτροπής. όπου συζητήθηκαν τι, συζητήθηκε τι ενέργειες αναλαμβάνει κάθε πλευρά και πώς μπορούμε καλύτερα να συνεργαστούμε. Είναι πολύ σημαντικό να βασιζόμαστε για τις ενέργειες μας αυτές σε κοινά στοιχεία. Το ΝΑΤΟ έδωσε ε, στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Επιτροπή, τη Στρατιωτική Επιτροπή του Συμβουλίου και επίσης έχουμε διαπιστώσει ότι οι ανάγκες στις στρατιωτικές που έχει εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτίζονται με αντίστοιχες ε, ανάγκες που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ με πολύ μικρές διαφορές. Αυτό είναι πολύ καλό, ε, μια πολύ καλή βάση για τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Μολενάρ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που τήρησαν το χρόνο ομιλίας ο λόγος στα μέλη της Επιτροπής μας, ξεκινώντας από τους συντονιστές και ο Ταξό. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω ονόματί μου και ονόματι της ομάδας μου, διότι έχει πιο θετικές από μένα η ομάδα μου. Θα μιλήσω προσωπικά, διότι είμαι πολύ λιγότερο ενθουσιώδης όσον αφορά τη στρατηγική κινητικότητα. Κατανοώ πολύ καλά το ότι θέλουμε να γίνει ένας παραλυσμός με τις τέσσερις βασικές ελευθερίες. Δεν μπορούμε μόνιμα όμως να ζητάμε οι στατιωτικοί να αντιμετωπίζονται με τις ιδιαιτερότητες ε, ε, που, έχει ο στατιωτικός τομέας και να κάνουμε όμως παραλληλισμό με άλλους τομείς όπως είναι η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και ανθρώπων. Ευτυχώς που οι στρατιωτικοί στην Ευρώπη δεν μετακινούνται όπως ο καθένας με θα ήταν ε, παρέκκληση να μπορούν οι στατιωτικοί να διέρχονται τα σύνορα έτσι, απλά, όπως τα αγαθά και υπηρεσίες, χωρίς ιδιαιτερότητα. Προσοχή, διότι αυτή η επιχειρηματολογία μπορεί να στραφεί κατά του σκοπού που θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Καταλαβαίνω όμως, παρόλα αυτά, τη χρησιμότητα να υπάρχουν πρωτόκολλα που επιτρέπουν τη διευκόλυνση της μετακινήσης προσωπικού υλικού αναφέρατε διάφορα θέματα και άειλα θέματα όπως είναι οι φόροι, οι διαδικασίες και έχετε απόλυτο δίκιο. Κατά την άποψή μου πρέπει να κάνουν προσπάθειες εκεί. Κατά τα λοιπά, αυτή η στρατηγική κινητικότητα όπως παρουσιάζεται, να το πω έτσι ειλικρινά, πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που ανήκει στο μεγάλο επίκαιρο θέμα. Κάθε 4-5 χρόνια η αμυντική κινητικότητα με την έννοια ε, του ε, όρου προσπαθεί να μειώσει τα γραφικατικά εμπόδια. Μερικά πράγματα δεν τα καταλαβαίνω. Για τη διευκόλυνση μετακινήσεων. Προς ζώνες ανάπτυξης στατευμάτων μιλάμε, ενεχόμενες ζώνες σύγκρουσης. Στο Ευρωπαϊκό Υπηρετικό Θέατρο βλέπουμε που θα μπορούσαν να είναι αυτές οι περιοχές, κυρίως προς την Ανατολική Ευρώπη. Οι περισσότερε χώρε κεντρική και ανατολική Ευρώπη έχουν προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ εδώ και 15 χρόνια. Βασικό στόχο του ΝΑΤΟ είναι η συλλογική άμυνα, άρθρο 5. Και 14 χρόνια μετά την προσχώρησή του λένε Α, δεν προβλέψαμε το προσωπικό και τα άρματα μάχη να μπορούν να αναπτυχθούν στα Ανατολικά αν υπάρχει πρόβλημα. Μα ποιον προσπαθούν να γελάσουν. Ανακάλυψαν το 2016 το πρόβλημα ότι είναι περίπλοκο να μετακινηθούν στρατεύματα και άρματα ε, στην Ανατολική Ευρώπη και δεν σκέφτηκαν τι, τι, τι, τι, τι κάνανε 14 χρόνια και θα την πληρώσει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση 6 δισεκατομμύρια έτσι. Στα καλά καθούμενα, να είμαστε σοβαροί. Δεν λέω ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν λέω ότι είναι ένα θέμα. Αλλά πόσο ελαφρά το αντιμετωπίσαμε το θέμα μέχρι τώρα. Και γιατί αυτό το θέμα τη εντικής κινητικότητας σαν μανιτάρι ξεφυτρώνει τώρα και είναι η προτεραιότητα, όλοι το συζητάνε και θέλουμε πολλά χρήματα και κουβεντιάζουμε, συζητάμε κλπ. Τι έγινε 14 χρόνια. Δεν υπήρχε ο χρόνο ε, να διαπιστωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα μετακίνηση αρμάτων μάχη και προσωπικού στην Ευρώπη. Ασχολούμεθα με αυτό τώρα, θα πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα γράψει με μεγάλη επιταγή. Θέλουμε περισσότερε λεπτομέρειε για αυτά τα διαβόητα προγράμματα. Εδώ και 10 χρόνια, εδώ, ήταν το pooling and sharing της μόδας να συναθίζονται οι πόροι. Κανεί δεν ξέρει τι έγινε. Ήταν το επίκαιρο θέμα, βάλτε χρήματα, συζήτηση κλπ. Ήταν τη μόδα. Comprehensive approach. Η σφαιρική προσέγγιση. Τώρα άλλο θέμα της μόδας, το military mobility, η στρατηγική κινητικότητα. Υπάρχουν θέματα βέβαια, υπάρχουν ζητήματα, τα αναφέρατε, αλλά πολιτικός πώς. Βέβαια το συζητάμε αυτό ακριβώς. Λέγατε πού πήγε ακριβώ. πολιτικά. Υπάρχει θέμα που πηγε όλο ο μηχανισμος Πώς συζητηση πω αυτο το θέμα τώρα ξεφυτρώνει. Με τέτοιο εύρο. Ενώ το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επί 14 χρόνια μπορούσαν να το επεξεργαστούν. Φαινόταν προφανέ. Και σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πληρώσει γι' αυτό. Αυτό που να το πω, μου φαίνεται κάπως χοντρό. Συγγνώμη που ήμουν έτσι επικριτικός υπερβάλλω πάντα, εκφράζομαι κάπως ζωηρά, αλλά θα ήθελα να το δούμε με ιστορικό βάθος αυτό το θέμα. Πώς καταλήξαμε σε αυτή την κατάσταση σήμερα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, από ό,τι μου είπαν ότι θα πρέπει να ε, ολοκληρώσουμε τη ζήτηση για το θέμα αυτό μέχρι τις 11.20. Έχω 9 ομιλητές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με να μην καθυστερήσουμε, να μην υπερβούμε το χρόνο μας. Επόμενος είναι ο κύριος Μίξα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ έχω πιο θετική στάση. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου. Συμφωνώ ότι καθυστερήσαμε. Θα έπρεπε να έχουμε αντιμετωπίσει τις δυσχέρες αυτές νωρίτερα. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Έτσι δεν είναι. Και δεν συμφωνώ με τον προηγούμενο μιλητή. Θεωρώ ότι δεν θα μας οδηγούσε ε, σε ανεξέλεγκτη κινητικότητα στρατιωτικών το να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ως πρώην Υπουργός Άμυνας δεν βλέπω καμία τέτοια απειλή. Αλλά για τις υποδομές. Θα πρέπει σε συνθήκες ειρήνης να μπορέσουμε να μετακινήσουμε στρατεύματα για λόγους ασκήσεων για λόγους εκπαίδευσης, αλλά και για αποστολές και στα πλαίσια της συνεργασίας με τον ΝΑΤΟ. Ξέρουμε ότι το ΝΑΤΟ δημιουργείται, δημιουργήθηκε για να υπάρξει προγραμματισμός και συλλογική άμυνα. Όλα αυτά σημαίνουν μετακινήσεις ενόπλων δυνάμεων, ενόπλων μονάδων από τη μία χώρα στην άλλη. Πρέπει να έχουμε και γενικά προγράμματα αλλά και πιο εξειδικευμένα προγράμματα για τη μετακίνηση μονάδων. Το προβλέπετε αυτό. για τα προγράμματα υποδομών ή είναι κάτι χωριστό. Είπε ότι σε γενικό επίπεδο είναι παρόμοιες οι απαιτήσει. Αλλά τα σχέδια του ΝΑΤΟ για έκτακτες παρεμβάσεις λαμβάνονται υπόψη στα προγράμματά σας για τη στρατιωτική κινητικότητα. Ο κύριος Άουστρα Κάγιο αργά παρά ποτέ και εγώ συμφωνώ. Άρα γιατί να μην προχωρήσουμε τώρα με τα προγράμματα στρατιωτικής κινητικότητας. Τα κριτήρια μα πρέπει να είναι τμήμα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, του κανονισμού για αυτά. Έτσι πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερα προγράμματα και έτσι και στρατιωτικά τμήματα θα μπορούν να μετακινούνται καλύτερα. Πείτε μου όμως, τι ποσοστό είναι η συμβολή των στρατιωτικών προγραμμάτων στην υλοποίηση των ε, άλλων προγραμμάτων υποδομών μεταφορών. Είναι 10, 15, 20%. Επίσης, σε τι βαθμό λαμβάνεται, υπόψη την πολυτροπικότητα των μεταφορών. Για να χρησιμοποιείτε όχι μόνο ε, φορτηγά και άλλα στρατιωτικά οχήματα, να χρησιμοποιείτε και τους σιδηροδρόμου. Είπατε στρατιωτική κινητικότητα η χερσαία. Με αυτήν έχετε ασχοληθεί. Δεν θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε και θαλάσσιες μεταφορές. Για να έχουμε μια συνολική στρατιωτική κινητικότητα. Η κυρία Ντεμιρέλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κάτι γενικό. Μας είπατε ότι υπάρχει αυτή η διτή χρήση. Όμως, στην έκθεση της, της κυρίας Μογκερίνη του περασμένου Ιουνίου αναφέρεται αυτή η διτή χρήση. Αλλά είναι σαφές ότι οι στρατιωτικές ανάγκες είναι το κύριο και οι στρατιωτικοί αποφασίζουν. Είναι λοιπόν σαφώς στρατιωτικό πρόγραμμα. Ξέρω ότι δεν σας αρέσει αυτό, αλλά αυτό είναι κατά των ευρωπαϊκών συνθήκων να αξιοποιούμε για στρατιωτικά προγράμματα ενωσιακούς πόρους. Είναι κατά του 41-2 τη συνθήκη Λισαβόνας. Παρ' όλα αυτά, Παρά αυτή την θεμεριώδη αντίθεσή μου, την συγκεκριμένη λοιπόν αντίθεση της ομάδας μου της αριστεράς, είπατε ότι θέλετε περισσότερη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ και ότι έγιναν συζητήσεις γι' αυτό. Πείτε μου λοιπόν, τι ρόλο παίζει το ΝΑΤΟ στα προγράμματά σας για τη στρατιωτική κινητικότητα. Και επειδή είμαι και Γερμανίδα, τι ρόλο παίζει το Γερμανικό Κέντρο Επιμελητίας. Πείτε μου. Επίσης, είπατε ότι η χρηματοδότηση αυτά τα 6,5 δις θα βγούνε από το προϋπολογισμό του συνδέοντας της Ευρώπη. Οπότε πείτε μου, αυτά τα 6,5 δις τι επιπτώσεις θα έχουν στην ε, πολιτική κινητικότητα, στις πολιτικές μεταφορές. Τι αρνητική επίπτωση θα έχουν. Διότι πρόκειται, ε, να το πω εντό εισαγωγικών, για παράνομη χρηματοδότηση στρατιωτικών προγραμμάτων. Ο κύριο Μπέργκ. Ευχαριστώ. Κύριε Κόλσον, με πολύ ενδιαφέρον άκουσα αυτά που είπατε στη Γερμανία μετά την επανένωση δεν επενδύθησαν αρκετά για προγράμματα διτής χρήσης. Το βλέπουμε κυρίως ε, στην υποδομή των σιδηροδρόμων. Δεν υπάρχει δυνατότητα στρατιωτικά οχήματα με ερπίστριες να χρησιμοποιούνται, να μπορούν να ανεβαίνουν σε σιδηροδρομικά βαγόνια. Δεν υπάρχουν κατάλληλες πλατφόρμες. Και επίσης η αυτοκινητόδρομή μας είναι σε άσχημη κατάσταση. Και αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατάσταση όπως την περιγράψατε. Και τα λαμβάνετε υπόψη σας γιατί και σε άλλα κρατημέλη είναι σημαντικά αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ κύριος Κρόσάι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν προσπαθώ να κάνω κάποιον διαχωρισμό ανάμεσα στη στρατιωτική και την πολιτική υποδομή. Στην πραγματικότητα, στον σύγχρονο κόσμο, οι υποδομέ μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε είναι στρατιωτικέ είτε είναι πολιτικέ. Για το ζήτημα τώρα της Ανατολικής Ευρώπης. Γνωρίζουμε ότι οι υποδομές πάσχουν. Είτε πρόκειται για πολιτικές υποδομές, είτε πρόκειται για στρατιωτικές. Αλλά επίσης και άλλα, άλλες υποδομές, όπως για παράδειγμα οι επικοινωνίες και ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που το έχουμε στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης από τη Βαλτική μέχρι τη Μεσόγειο. Το ερώτημα λοιπόν είναι, δεν πρέπει να κάνουμε κάτι για να βελτιώσουμε αυτές τις κατά κύριο λόγο πολιτικές υποδομές και να τις βελτιώσουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορέσει και ο στρατός να τις χρησιμοποιήσει αν χρειαστεί, γιατί διαφορετικά οι στρατιωτικοί θα πρέπει να κάνουν το δικό του σχεδιασμό. Ε, κάποια στιγμή την άνοιξη του 2015 νομίζω ε, υπολογίστηκε ότι θα χρειαζόταν ένας μήνας για να γίνουν κινήσεις 40.000, ε, ε, μιας μονάδας 40.000, ε, δυναμικής 40.000. Και αυτό είναι πολιτικό πρόβλημα. Επομένως δεν θα πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές πολιτικής χρήσης, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουμε και τη στρατιωτική χρήση. Γιατί γνωρίζουμε ότι οι υποδομές είναι διπλής χρήσης. Δεν πρόκειται δηλαδή να σπαταλήσουμε χρήματα για κάτι που δεν θα βοηθήσει και τους πολίτες. Δεν θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε, να, να βελτιώσουμε τη διασύνδεση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως εξυπηρετώντας την πολιτική χρήση, αλλά και την στρατιωτική. Εγώ έτσι βλέπω το θέμα. Το ζήτημα λοιπόν είναι πώ βελτιώνουμε τι υποδομέ μα κυρίω για του πολίτε τη Ένωση και δευτεραβόντω και για τη στρατιωτική χρήση του. Κύριο Πίτα. Ευχαριστώ. Για άλλε τι πληροφορίε που μα δώσατε, δεν είναι καινούριο το θέμα. Εγώ το γνωρίζω ήδη από τότε που εργαζόμουν στο, στο στρατό Μία από τις ασκήσεις που είχαμε είναι πώς θα μετακινούνταν τα θωρακισμένα από την Αμβέρσα στη Γερμανία. σήμερα με τη Γερμανία. Το ζήτημα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Κάτι ενδιαφέρον που αναφέρατε είναι ακριβώς αυτή η διπλή χρήση. Και Είπατε ότι τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες θα γίνουν διάφορες συναντήσεις για τον, να καθοριστεί ακριβώς τι εννοούμε για διπλή χρήση και πώς ε, αυτό επηρεάζει το σχεδιασμό μας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε να ενημερωθούμε όταν τελικά αυτή η συζήτηση κλείσει. Δεύτερον, έχουν τεθεί κάποιες προτεραιότητες σε σχέση με τη διπλή χρήση, γιατί φαντάζομαι ότι το ζήτημα θα ενδιαφέρει πολλά κράτη-μέλη και ότι κατά πάσα πιθανότητα θα προταθούν περισσότερα έργα από ότι ο διαθέσιμος προπολογισμό θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει. Έχουν τεθεί προτεραιότητες και ποιος θα λάβει τις αποφάσεις τελικά. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Γιούρη και έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Οι εγκληματίες είναι πιο αποτελεσματικοί από την συνεργασία στην Ευρώπη για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Γιατί έχουμε αυτά τα σύνορα, τα οποία εμείς ήδη έχουμε ε, δημιουργήσει, όλα αυτά τα εμπόδια που μας παρέγραψε ο κύριος Κολσό, δεσμολογικά, φορολογικά. Και αυτό είναι λυπηρό αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο σημαντικό είναι και ο στρατός όπως οι γιατροί, η αστυνομία να έχει τη δυνατότητα να δρά διασυνοριακά. Το πρόβλημα είναι κυρίως στην Ανατολή. Στρατηγικής ε, φύσεως προβλήματα έχουμε στην Ανατολή και στον Βορρά. Και βεβαίω υπάρχει και το ζήτημα ε, μια κρίση στον Ατλαντικό, αλλά αυτό είναι γενικότερο. Εάν η κίνηση του στρατιωτικού εξοπλισμού γίνει θαλάσσης, αυτό είναι πολύ περίπλοκο και χρονοβόρο. Επομένως, η καλύτερη ε, ε, κινητικότητα μπορούμε να την έχουμε με τη χρήση των σιδηροδρόμων. για ιστορικούς λόγους υπάρχουν αυτά τα προβλήματα ε, και έχουμε εμείς το πρόβλημα της Ιβηρικής Χερσονήσου που δεν είναι σωστά συνδεδεμένη ε, με την υπόλοιπη πυρωτική Ευρώπη. Πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αξιοπρεπή στρατιωτική κινητικότητα προς την Ιβυρική Χερσόνησο και από αυτήν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στρατιωτική κινητικότητα είναι ουσιαστικό στοιχείο της δυνατότητας των στρατιωτικών μας δυνάμεων να ανταποκρίνονται σε κρίσεις. Πολλές στρατιωτικές ασκήσεις δεν ε, κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν στη Ρουμανία εξαιτίας της κατάστασης των υποδομών μας. Ε, Ιδίω όταν σε αυτέ τι ασκήσει συμμετείχαν αμερικανικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Το 2004 είχαμε το ένα περιστατικό ενό τρένου που ε, μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό, το οποίο ε, μπλοκαρίστηκε σε έναν μικρό σταθμό τρένων για πάνω από 20 ώρες μέχρι να λυθεί ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα. Δεν έχουμε πια τέτοιου είδους προβλήματα, έχουμε όμως ένα διαφορετικό πρόβλημα. Το εξή. Μιλούμε για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού. Ε, και τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και μέλη του ΝΑΤΟ πρόβλημα που εγώ λοιπόν εντοπίζω και το είχα εντοπίσει και παλαιότερα που ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής είναι ότι πρόκειται περί του ίδιου εξοπλισμού, δηλαδή μεταφέρουμε τον εξοπλισμό τον οποίο τον είχαμε διαθέσιμο για το ΝΑΤΟ, για τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ και τον σκεφτόμαστε να τον μεταφέρουμε αυτόν τον εξοπλισμό και αυτούς τους πόρους προς χρήση από την, ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν σκοπεύει κανείς να έχει δύο διαφορετικές ε, εξοπλισμό ή δυνατότητες. Και αναρωτιέμαι αν αυτό είναι ρεαλιστικό. Μέχρι στιγμής το ΝΑΤΟ έχει αποδείξει την αποτρεπτική του ισχύ έχει αποδείξει ότι αποτρέπει οποιονδήποτε από την ιδέα ή την πιθανότητα να ξεκινήσει μια σύγκρουση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μέχρι και στο έδαφος της Ρωσίας και το λέω αυτό γνωρίζοντας τι συμβαίνει στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Γνωρίζω ότι η Ρωσία, γνωρίζουμε ότι η Ρωσία δεν έχει τολμήσει να απειλήσει κανένα κράτος στη δυτική στο δυτικό ημισφαίριο. Επομένω, το ερώτημα είναι γιατί χρειάζεται ένας ευρωπαϊκός στρατός και πώς θα το δικαιολογήσουμε αυτό στους πολίτες μας. Μετά τη ρωσική κατάληψη της Κρυμαίας και της Ανατολικής Ουκρανίας, τι συνέβη. Έγινε μια σύνοδος κορυφής στην Ουαλία και το συμπέρασμα ήταν ότι ουσιαστικά θα διευκολύνουμε τη μεταφορά ε, στρατευμάτων και εξοπλισμού κατά κύριο λόγο αμερικανικού και αμερικανικών στα ανατολικά σύνορα. Το ΝΑΤΟ λαμβάνει υπόψη του τους σημαντικούς κινδύνους που υπάρχουν στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. το ζήτημα της ασφάλειας μπορεί να το δει κανείς διαφορετικά ανάλογα με την ε, οπτική που επιλέγει. Κατά την άποψή μου, την ειρήνη μπορούμε να τη διασφαλίνουμε με την αποτρεπτική ε, ισχύ του ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ κύριε Μπασέσκου. Τώρα στο πάνελ να στραφώ. Αντίθετη σειρά θα πρότεινα. Παρακαλώ προσπαθήστε να είστε όσο πιο λακωνική μπορείτε, περίπου ένα τετράλεπτο ο καθένας, για να προλάβουμε. Ο κ. έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομος. Ευχαριστώ για τα σχόλια, ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις. Σημαντικότατο αυτό το πρόγραμμα, άρα χρήζει της δέουσας προσοχής και ανάλυσης. Αυτό το έργο που κάνουμε, η στατιωτική κινητικότητα, ανταποκρίνεται στι ανάγκε των κρατών μελών. Αυτό τελικά καθοδηγεί τις εργασίες μας. Όπως προανέφερα, βασιζόμαστε στην πραγματική εμπειρία των ενόπλων δυνάμεων της Ευρώπης. Όχι μόνο σε στιγμές κρίσης, αλλά όταν ετοιμάζονται για ασκήσει, ε, διμερεί ή πολυμερεί ασκήσει πρέπει να μεταφέρονται στα τεύματα διασυνοριακά στην Ευρώπη. Και για να διευκολυνθεί αυτό και να εξομαλυνθεί, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτό που θέσαμε σαν στόχο. Δεν είναι ότι θα αναλάβει ρόλο συλλογική άμυνα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΝΑΤΟ το κάνει αυτό, είναι σαφέ. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίνεται στι αμυντικέ ανάγκε των μελών τη. Αυτό είναι το βασικό που θα ήθελα να διευκρινίσω. Κάποια άλλα στοιχεία αναφέρθηκαν στη συζήτηση δεν υπάρχει ε, πολιτική, ή στατιωτική υποδομή, εκτός αν μιλάμε στατιωτικέ ε, βάσεις που είναι στατιωτική υποδομή. Για τις μεταφορές έχουμε ένα ενίο δίκτυο, πρωταρχικά προς πολιτική χρήση, αλλά ίσως σε καιρούς ειρήνης ή σε περίπτωση κρίσης οι στατιωτικοί πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτές οι υποδομές. Αυτό είναι το πλαίσιο της συζήτηση. σωστή προσέγγιση θα αφήσω του άλλου συναδέλφου να αναφερθούν στα θέματα θέσεως προτεραιοτήτων κλπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Πιστεύω ότι οι συνάδελφοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα θέλουν να απαντήσουν περισσότερο να έχουν τον χρόνο. Ο φορέας μας έχει ρόλο υποστήριξη των δράσεων, στατιωτικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένους οριοθετημένους τομείς, διαδικασίες, εναρμόνιση στοιχείων για τη μείωση του διοικητικού άχθους, Παρεμβαίνουμε με ρόλο υποστηρικτικό κατόπιν αιτήματο των κρατών μελών στα πλαίσια του Action Plan. Έτσι αντιλαμβάνομαι τι ερωτήσει σα, αλλά σαν εκπρόσωπο του φορέα μου δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά που θέσατε σήμερα. Ευχαριστώ, κύριο Κόλσον. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Οι επενδύσεις πού θα γίνουν παντού, παντού στην Ευρώπη. Μετά την ερώτηση του κυρίου ε, ε, του Ισπανού Ευρωβουλευτού θα αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Ακόμα και αν μπορούμε να παραδεχθούμε ότι οι περιορισμοί ή οι απειλές μάλλον προέρχονται εξ Ανατολών, θα πρέπει εν πάση περιπτώσει να περάσουμε στρατεύματα καμιά φορά από την... να μεταφέρουμε τα στρατεύματα από την Νότια Ισπανία. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτήσει ένα συγκεκριμένο μέσο Ευρώπης και όχι αλλού όλη η Ευρώπη σύμφωνα με τις ανάγκες στρατιωτικής κινητικότητας θα έχει πρόσβαση σε αυτή τη χρηματοδότηση. Γιατί τώρα. Όπως είπα και συνάδελφοι, διότι τα κράτη-μέλη μας το ζήτησαν. Ίσως και πιο απλά, διότι κάποιες απειλές που αντιμετωπίζουμε είτε στην Ουκρανία είτε τρομοκρατικές απειλές είναι γεγονότα πρόσφατα και επιβάλλεται τώρα να βρεθεί η λύση. Περισσότερο είναι πιο ε, με μεγαλύτερη οξύτητα τίθεται τα προβλήματα από ό,τι εδώ και 15 χρόνια. Τώρα, αν πρόκειται για αποτυχία του ΝΑΤΟ, σίγουρα όχι. Όχι, αν πρόκειται για μια επιταγή που δίνουμε στο ΝΑΤΟ, καθόλου. Το ΝΑΤΟ χρηματοδοτεί αποκλειστικά στατιωτικές υποδομές. Αυτό είναι ο ρόλος του ΝΑΤΟ. Ο στόχος του μηχανισμού που προτείνεται είναι χρηματοδότηση ε, πολιτικών ε, υποδομών, υποδομών για πολιτική χρήση μέχρι το επίπεδο και το βαθμό που θα είναι χρήσιμες υποδομές για πολιτική χρήση. Στο βαθμό που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στατικοί από στατιωτικού αυτέ οι υποδομέ. Τα περισσότερα μεταφορικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται από του στατιωτικού ε, είναι υποδομέ για την πολιτική χρήση. Ναι, η πολυτροπικότητα των μεταφορών αποτελεί ένα τμήμα των υποδομών που θα χρηματοδοτηθούν. Εξάλλου δεν θέλουμε να αποκλείσουμε οποιοδήποτε μεταφορικό τρόπο. Κάθε τρόποι μεταφοράς που όλοι οι τρόποι χρησιμοποιούνται τακτικά από τους στρατιωτικούς, κυρίως το δικό δίκτυο και οι σιδηρόδρομοι, είναι σημαντικοί τομής, αλλά όλοι οι τρόποι μεταφοράς θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Οπότε και τα κριτήρια διπλής χρήσης καταρτίζονται για όλους τους τρόπους μεταφορών. Αυτό καλύπτει και τις θαλάσσιες μεταφορές. Δεν θα υπάρξει καμία χρηματοδότηση από το μηχανισμό για τις μεταφορές στην Ευρώπη, αν δείτε το πλαίσιο το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, ο προπολογισμό του μηχανισμού για τι διασυνδέσει, για τι μεταφορέ στην Ευρώπη ε, παραμένει στο ίδιο επίπεδο, μετάβλητο. Συμπληρωματικό κονδύλι που ανήκει στο κεφάλαιο άμυνα και ασφάλεια είναι αυτό που προβλέπεται για τη στρατιωτική κινητικότητα. Και αυτό το συμπληρωματικό κονδύλι θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις που θα είναι χρήσιμες για θέματα πολιτικής χρήσεως δεν υπάρχει μετακίνηση, απορρόφηση από, από μία χρήση για άλλη, αλλά συμπροματικό ποσό για αισθητική χρήση που θα είναι και χρήσιμο και για τον πολιτικό. Το υπόλοιπο του, του μηχανισμού για την κινητικότητα στην Ευρώπη ε, παραμένει αμετάβλητο. Δεν θα απορροφηθούν πόροι, δεν θα αφαιρεθούν πόροι από το ΣΕΦ για να πάνε για αυτή τη χρήση που συζητάμε τώρα. Άρα δεν επιβαρύνονται οι κλασικές ε, ε, τακτικές δραστηριότητες ε, του όλου μηχανισμού κινητικότητας διασυνδεσιμότητας Ευρώπης. Πώς θα λειτουργήσει αυτό. Όπως λειτουργεί ο μηχανισμός για τη διασυνδεσιμότητα στην Ευρώπη. Υπάρχουν προτεραιότητες διαγωνισμοί για υποβολή προτάσεων. Αυτές οι προτεραιότητες ε, είναι διαφανείς, δημοσιοποιούνται. Τα κράτη-μέλη μπορούν να προτείνουν διάφορα προγράμματα και έργα και αυτά τα προγράμματα μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης σε, μέχρι επίπεδο 50% διότι αυτό έχει αποφασιστεί από τους συνομοθέτες. Ναι, σίγουρα είναι μια προτεραιότητα και για τον πολιτικό και στατιωτικό τομέα να φροντίσουμε ούτως ώστε ε, η διαφορά, να, το εύρος των, από τις ράγες στην ε, Ιβηρική ε, Ήπειρο να ταυτιστεί και με το εύρος το, από τις ράγες που υπάρχει και στις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ιδού λοιπόν αυτά κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστούμε τους τρεις ομιλητές μας. Ευχαριστώ που ήσασταν από το πρωί μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Μα να επανέλθω στην ερώτηση. Σας παρακαλώ... Σας παρακαλώ, ε, έχουμε μεγάλη καθυστέρηση, διμερός παρακαλώ. Μα δεν έλαβα μια πολύ σημαντική απάντηση. Από πού θα είναι τα στρατεύματα. Από πού θα αφαιρεθεί αυτή η δυνατότητα, από το ΝΑΤΟ ή από αλλού. Γιατί δεν μου αρκεί η απάντηση ότι αυτό είναι αίτημα των κρατών μελών. Η πρωτοβουλία δεν σκοπεύει να επιβάλλει στρατιωτικές κινήσεις στα κράτη-μέλη η πρωτοβουλία θα επιτρέψει τα κρατη στα κράτη-μέλη, στις ένοπλες δυνάμεις τους, να μετακινούνται πιο εύκολα. Ωραία, καλά κάνα μια εξαίρεση. Ευχαριστούμε τους ομιλητές. Λοιπόν, τώρα χρειαζόμαστε και μια σύντομη διακοπή γιατί δεν έχει έρθει ο επόμενος ομιλητής μας. Άρα θα μπορούσαμε να έχουμε συνεχίσει τη συζήτηση. Αλλά μόλις τώρα μου είπαν ότι λείπει ο επόμενος ομιλητής. Πέντε λεπτά διακοπή. Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, Λοιπόν, σημείο 5 τη ημερήσια διάταξη. Ανταλλαγή απόψεων για τι ε, συντονισμένε θαλάσσιε παρουσίε. Έχουμε δύο προσκεκλημένου. Του καλωσορίζω. Όταν είναι ο κύριο Ζακ Φαντά, που είναι τμήματάρχη για την, ε, τον ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και τη σταθεροποίηση έχει συμβάλει στην ε, επεξεργασία του όρου αυτού της ε, συντονισμένης θαλάσσιας παρουσίας. Μας ενδιαφέρουν πολλά αυτά που θα μας πείτε. Είμαι βέβαια. Και καλωσορίζω και τον ε, λοχαγό Hans Huygen που είναι στην διεύθυνση του στρατιωτικού σχεδιασμού και αξιολόγηση. Λοιπόν, παρακαλώ, 10 λεπτά ο καθένας. Και μετά θα κάνουμε ανταλλαγή απόψεων. Παρακαλώ κύριε Φαντά, εσείς. Ευχαριστώ. Πάντα χαρά να είμαι εδώ μαζί σα για να σα εξηγήσω τι κάνουμε για τις συντονισμένες θαλάσσιες ε, παρουσίες. Λέγομαι Ζακ Φαντά, είμαι τμήματάρχης στο λεγόμενο τμήμα ISP. Η θάλασσα είναι επίκεντρο γεωστρατηγικής αντιπαράθεσης παγκοσμία. Τα κράτη-μέλη της Ένωσης τακτικά αναπτύσσουν ε, θαλάσσια μέσα αρκετά σημαντικά παντού στον κόσμο. Το σχέδιο δράσης για τη στρατηγική θαλάσσιας ασφάλεια της Ένωσης αναθεωρήθηκε το 2018 με βάση την παγκόσμια στρατηγική της Ένωσης. Η Ένωση λοιπόν θέλει να παίξει σημαντικότερο ρόλο στη θαλάσσια ασφάλεια, στην ασφάλεια των θαλασσών. Τα απορίσματα του Συμβουλίου για την Ασφάλεια και την Άμυνα που εγκρίθηκαν τον περασμένο Ιούνιο επίσης καλούν να γίνει ένα στρατηγικός προβληματισμός για την παγκόσμια στρατηγική παρουσία της Ένωσης. Γι' αυτό ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία. Πώς θα συντονίσουμε καλύτερα την παρουσία των κρατών μελών στις θάλασσε εθελοντικά βεβαίω. ούτω ώστε να αποφεληθούμε περισσότερο πολιτικά και λειτουργικά. Η Ένωση με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να ενισχύσει την ασφάλεια των θαλασσών εκεί που υπάρχουν παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες που προκαλούν κινδύνους για τις θαλάσσιες μεταφορές. Αλλά όχι μόνο για τι μεταφορές. Πέρα από αυτό το στόχο, που είναι ο κύριος στόχος, έτσι θα παίξουμε καταλητικό ρόλο για την παγκόσμια δράση τη Ένωσης. Διότι μπορούμε να ενισχύσουμε το ρόλο μας ως πλατφόρμα που θα συμβάλλει στην ασφάλεια των θαλασσών, βέλτιστοποιώντα τι δυνατότητε των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Η έννοια συντονισμένη στρατηγική παρουσία είναι το νέο εργαλείο για να το κάνουμε αυτό. Αυτή η έννοια παρουσιάστηκε τον περασμένο Ιούλιο, συζητήθηκε στο Ελσίνκι, στο Συμβούλιο των Υπουργών και ενεκρίθη από τα κράτη-μέλη για να ε, δοκιμαστεί στον κόλπο της Γουινέας. Είναι από κάτω προς τα πάνω στρατηγική, προσεκτική και ρεαλιστική για να έχουμε ένα ρωμαλαίο ανθεκτικό εργαλείο. Βασιζόμαστε σε θελούσιες σύμβολες των κρατών μελών και τα μέσα παραμένουν υπό εθνική διοίκηση. Η συντονισμένη θαλάσσια παρουσία είναι ένα νέο μέσο, ευέλικτο, βασίζεται στα διδάγματα των ε, θαλασσίων επιχειρήσεων της Ένωσης. Συγκεκριμένα της Αταλάντα στον Ινδικό ωκεανό και της ε, Σοφία στη Μεσόγειο. Έχουμε και τις ε, παράλληλες πρωτοβουλίες όπως είναι το κέντρο για την θαλάσσια ασφάλεια, το ΜΣΟΑ ή και άλλους μηχανισμούς συντονισμού, όπως το ΣΕΙΤ. Βασίζεται και σε πιο πρόσφατες εμπειρίες, όπως ε, η παρουσία μιας γαλλικής ε, φρεγάτας ε, που αγκυροβόλησε στη, στο Μουμπάι. Έτσι ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στον τομέα αυτό με την Κίνα. Οι τρεις κύριοι στόχοι συνδέονται στενά. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να αυξήσουμε την στρατηγική και λειτουργική παρουσία της Ένωσης σε συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Δεύτερον, να αυξήσουμε την κοινή γνώση μας για την κατάσταση των θαλασσών. Και τρίτον, να αυξήσουμε τη δράση μας για να διευκολύνουμε ορισμένες δράσεις σε συνεργασία με τους εταίρους μας. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να καθορίσουμε τις περιοχές ε, που μας ενδιαφέρουν στις θάλασσες, το πιο ψηλό πολιτικό επίπεδο, υποθέτω επίπεδο Συμβουλίου. Έτσι τα κρατη θα μπορούν εθελούσια να προτείνουν σκάφη για να εφαρμόσουν τους στόχους. Για να υπάρχει καλύτερη γνώση των θαλασσών, πρέπει να συλλέξουμε και να αναλύσουμε πληροφορίες με βάση τη χρήση των σκαφών και άλλων μέσων που δίνουν τα κράτη-μέλη ούτως ώστε να ε, βελτιώσουμε και τη στρατηγική μας. Η ανάγκη να έχουμε στρατηγικό συντονισμό όπου θα καταλήγουν όλες οι αναλύσεις μας καθώς και η καθοδήγηση των ε, ενεργειών μας έχουν ήδη εντοπιστεί. Ε, χρειάστηκε λοιπόν να αποφασίσουμε να κάνουμε στον κόλπο της Γουινέας μια δοκιμή των μεθόδων μας, στηρίζοντας τη στρατηγική της Ένωσης για να αναπτύξουμε περαιτέρω την αρχιτεκτονική του Γιαουντέ. Το σχέδιο εφαρμογή είναι υπό Θα προταθεί στα κράτη-μέλη προ έγκριση πριν από το τέλο του χρόνου. Παράλληλα, θα συζητήσουμε τη μελλοντική χρήση του εργαλείου αυτού μέσω μιας διαδικασίας καθορισμού των θαλασσίων περιοχών που μας ενδιαφέρουν. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Χόχινς. Δεν έχω να προσθέσω και πολλά. Πέρα από το ότι μέσω του, στο στρατιωτικό επιτελείο παρέχουμε την σχετική γνώση που χρειάζεται για τον ολοκληρωσμένο σχεδιασμό και εμείς συνεισφέρουμε τη γνώση των θαλασσών, εγώ και οι συναδελφοί μου. Από τις εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει από τη συμμετοχή μας στις διάφορες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και από τα διδάγματα που αντλούμε από τις επιχειρήσεις των κρατών μελών. συνεχίζεται ε, η δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια ε, προσέγγιση που πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Αυτά από την πλευρά μου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Αμυντική Στρατηγική ρεαλιστικά μιλώντας, βασίζεται πρώτα απ' όλα στα εθνικά συμφέροντα και μετά, εάν είναι εφικτή συνεργασία, την εφαρμόζουμε. Αλλά η παρουσία στην θάλασσα ε, του ναυτικού είναι πρώτα απ' όλα μια παρουσία εθνική και μετά ευρωπαϊκή. Έχουμε να αντιμετωπίζουμε παγκόσμιες προκλήσεις. Όμως εμείς συνεχίζουμε να έχουμε μια πολιτική κατά κύριο λόγο εθνική. Πέρα λοιπόν από την επιθυμία την οποία έχουμε εκφράσει όλοι. Έχουμε να αντιμετωπίσει ε, απειλές τρομοκρατικές εξαιρετικά περίπλοκες που χρειάζονται για να αντιμετωπιστούν συντονισμό, όπως για παράδειγμα στην περιοχή της Σομαλίας. Και εκεί στην περιοχή της Σομαλίας η παρουσία είναι κατά κύριο λόγο εθνική, είναι βρετανική και γαλλική από πλευράς Ευρώπης. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργεί προς όφελος των ε, συμφερόντων κάθε κράτους μέλους, μπορεί να οδηγεί σε δυσλειτουργίες όσον αφορά την ευρωπαϊκή παρουσία. Ευχαριστούμε κύριο Πέτρας. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε και για την ενημέρωση ευχαριστώ. Πιστεύω ότι είναι θετική πρωτοβουλία αυτός, αυτή η προσπάθεια συντονισμού. Θα ήθελα να με ενημερώσετε εάν υπάρχει συνεργασία με το ΝΑΤΟ για τα θέματα αυτά. Υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, ποια είναι η φύση της ε, σχέσης μας με το ΝΑΤΟ, τις σχέσεις της πρωτοβουλίας της δικής μας με αυτό που κάνει το, ή δεν κάνει το ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ, θα δώσω το λόγο στους ομιλητέ μας. Ευχαριστώ τους δύο μιλητές για τις ερωτήσεις τους. Για το ζήτημα του ΝΑΤΟ και φαντάζομαι και ο συνάδελφος θα δώσει περισσότερες πληροφορίες η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ στον τομέα του, ναυτικού είναι εξαιρετική και το βλέπουμε ε, ήδη στις διάφορες κοινέ επιχειρήσεις. Βεβαίως, θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον η συνεργασία μας με τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, αυτή τη στιγμή γίνεται κατά περίπτωση και αναζώνει. με βάση μια πολύ βασική αρχή να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις. Όπως σας έλεγα λοιπόν και πριν, αυτή τη στιγμή ε, κάνουμε διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη για να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και στο μέλλον επί τη βάση των εμπειριών που θα αποκτήσουμε με την επιχείρησή μας, με την παρουσία, παρουσία μας στον κόλπο της Γουινέας. Ε, αν προσθέσω κι εγώ για την συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, όπως ήδη αναφέρθηκε. Ε, υπάρχει ε, παρελθόν σε αυτή τη συνεργασία και ήταν πολύ επικοδομητική επί πολλά χρόνια. Αυτό λοιπόν που έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά στο κέρας της Αφρικής και στη Γουινέα δεν νομίζω, δεν βλέπω γιατί να μην λειτουργήσει και σε αυτήν την περίπτωση εδώ πρόκειται εξάλλου για συντονισμό, δεν πρόκειται για επιχείρηση. Όμως, μιας και ε, βρισκόμαστε σε αρχική φάση, έχουμε προγραμματίσει να γίνουν τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και όπως είπε ο κ. Φχαντά, συνεργαζόμαστε και με τα κράτη-μέλη, πρώτα απ' όλα αυτή είναι η κυρία μας προτεραιότητα, αλλά επίσης και με τον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, πλειοκτήτες ε, και αντίστοιχες ε, επιχειρήσεις του κλάδου γιατί είναι εκείνοι οι οποίοι πλήττονται από ε, τα, προβλήματα αυτά στη θάλασσα. Θα δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με τον ΝΑΤΟ λαμβάνοντας βεβαίω υπόψη μας το γεγονό ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν, έχουν μία δύναμη την οποία αναπτύσσουν και επί τη βάση των απαιτήσεων και του ενός οργανισμού και του άλλου. Και του ΝΑΤΟ δηλαδή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έρχομαι τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Η συμμετοχή θα είναι θελοντική. Η αξιοποίηση είτε σκαφών, είτε αεροσκαφών, είτε ομάδων θα γίνεται ε, κατόπιν αιτήματο, αλλά θα πρέπει να είναι ε, έτοιμε αυτές οι μονάδες ε, να αναπτυχθούν. Θα πρέπει να είναι έτοιμοι επιχειρησιακά και κάθε κράτος θα τις προσφέρει σε θελοντική βάση στη, μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά όπως διευκρινίστηκε, η ε, ο συντονισμός θα γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμένουν ε, όσον αφορά τις συντολές που θα λαμβάνουν υπό έλεγχο εθνικό. Κύριε Σφραγκά, σας ευχαριστώ πολύ. Η ερώτηση που θέσατε καλύπτει και κάτι γενικότερο από αυτό που συζητούμε σήμερα για την θαλάσσια παρουσία. Αλλά αυτό που περιγράψατε συνεισφέρει και στο δικό μας προβληματισμό. Βεβαίως έχουμε πιο σημαντική θαλάσσια παρουσία στις ε, περιοχές που αναφέρατε. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες ζώνες που πιθανώς να μας ενδιαφέρουν, όπως για παράδειγμα η ρεκτική. Μέχρι τώρα έχουμε επιλέξει να εστιάσουμε στον κόρπο της Γουινέας. Και βεβαίως το ζήτημα θα τεθεί κάποια στιγμή πολιτικά σε ποιε γεωγραφικές περιοχές θα εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία του συντονισμού. Το γεγονό ότι πρόκειται για μια εθελοντική ανταλλαγή πληροφοριών και μια ενίσχυση της παρουσίας ε, και της ε, εφαρμογή, προς το στόχο της εφαρμογής της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι θετικό αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι ίσως κάποια στιγμή υπάρξουν και δυσκολίες γιατί οι διαθέσιμοι πόροι, οι διαθέσιμες δυνάμεις είναι ε, περιορισμένες. Αλλά βέβαια αυτό το πρόβλημα φαντάζομαι θα αργήσει, θα το αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Ελπίζω να απάντησα στο ερώτημά σας. Κύριε Νάτ. Ερώτηση πρακτική, πρακτικού χαρακτήρα. Πώς είναι η συνεργασία μεταξύ της αποστολής της Ένωσης στον κόλπο της ε, Γουινέας και των αρχών της Νιγηρίας, γιατί οι πειρατές έχουν τη βάση τους στην Νιγηρία. Και ξέρουμε νομίζω όλοι πόσο διεφθαρμένη είναι η δημόσια διοίκηση εκεί. Αν δεν είχαν λιμάνι να βρουν οι πειρατές, δεν θα ε, μπορούσαν να κάνουν αυτό που κάνουν. Επομένως, ποια είναι η με τις αρχές ε, της ε, Νιγηρίας. Γιατί αν δεν κερδίσουμε το παιχνίδι και στην ξηρά, ε, είμαστε χαμένοι. Τεράστιο ερώτημα. Εκεί σχαντέμισα, Δεν είναι το πρόβλημα. Πώς αντιμετωπίζουμε τη θαλάσσια πειρατεία, αν η χώρα εντό αγωγικών, από, εισαγωγικών, από εκεί που προέρχονται οι πειρατές, δεν συνεργάζεται ή δεν μας δίνει τα μέσα για να κινηθούμε. Ε, στο κέρας Αφρικής ε, μπορούμε να συγκρίνουμε αυτό που κάνουν στις αρχές της Σομαλίας και με αυτά που συμβαίνουν στον κόλπο της Γουινέας. Κοιτάξτε, προσπαθούμε να βρούμε απάντηση. Μαζί με τους εταίρους προσπαθούμε να δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η αρχή Το κονσέπτ δημιουργούμε, ε, είναι ένα hot spot εκεί πέρα στον αυτή πειρατεία. Έχουμε κάποιους περιορισμούς στον αυτή τη και κυκλοφορία. Έχουμε διάφορους μοχλούς πίεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για τις επαφές με τις τοπικές αρχές μέσω αντιπροσωπιών, μέσω κρατών μελών, μέσω πρωτοβουλίων των εταίρων μας. Και υπάρχουν τέτοιες με τρίτες χώρες που έχουν συμφέροντα στην περιοχή. Το ότι εξετάζουμε τι μπορεί να γίνει στον κόλπο της Γουινέας είναι μια πρώτη καλή προσέγγιση για να δούμε τι μέσα και μοχλούς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να έχουμε συγκεκριμένη δράση που δρομολογήσουμε. Ούτως ώστε να μειώσουμε πρώτης τις συνέπειες που περιγράψατε. Ευχαριστώ κύριε Φάλα. Κύριε να προσθέσω κάτι. Θα χρησιμοποιήσουμε ε, εθνικά μέσα υπό εθνικό έλεγχο και εξαρτάται από τα κράτη-μέλη να καθορίσουν το με ποιες χώρες θα συνεργαστούν καταρχάς σε στενό συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ε, τον πρώτο λόγο έχουν τα κράτη-μέλη και γι' αυτό Προσπαθούν να, προσπαθούμε να πετύχουμε αμοιβαίο όφελο καταρχάς και για το κάτω μέλο που δίνει το μέσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα συμμετάσχουν χώρες όπως η Νιγηρία. Αυτό δεν γίνεται μόνο σε εθνικό επίπεδο, μέσω περιφερειακού επίπεδου, με οργανώσει όπως είναι η Αφρικανική Ένωση και μέσω Τσέκοβας, που είναι ισχυρό περιφερειακό φορέα που μπορεί να έχει μεγαλύτερη επιρροή όσον αφορά την κακή συμπεριφορά ούτως υπήν αυτών των κρατών. Ο κύριος Πίτερς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Άλλη μια σύντομη ερώτηση. Όταν συμβεί το Brexit, κάτι που απέφχονται όλοι, όταν υπάρξει Brexit, ποια θα είναι η συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και της πρωτοβουλία που συζητάμε. Καλή ερώτηση, λέει Πρόεδρος. Κύριε Σχάτε. Έξοχη ερώτηση. Δεν νομίζω ότι έχω κάθε όλες τις απαντήσεις. Να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Να ξέρουμε, ας πούμε, τι χορό θα χορεύσουμε τους Βρετανούς συναδέλφους. Έγιναν προτάσεις για ενδεχόμενη συνεργασία με τους Βρετανούς θα έχουμε συνεργασία όπως με τρίτη χώρα ή κάτι άλλο. Το ιδεώδες θα ήταν να παραμείνουν στην οικογένειά μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά κανείς δεν έχει σήμερα κρυστάλλινη σφαίρα για να γνωρίζει ακριβώς πώς θα γίνουν όλα αυτά. Ελπίζουμε τελικά η κοινή λογική να επικρατήσει, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ και τους δύο σας. Νομίζω ότι θα συνεχιστούν προγράμματα αυτού του είδους. Ευχαριστώ πολύ συνεργασία. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις. Πολύ καλές ερωτήσεις. Τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξη 6. Παρουσίαση της μελέτες για το δίκτυο της Νορμανδίας, αξιολόγηση των απειλών κατά της ε, ειρήνης. Θα αφήσουμε πρώτα τους φιλοξενούμενους μας να αποχωρήσουν. Let's uh, συνεχίσουμε. Από τον Ιούνιο του 2018 διεξάγεται συνεδρίαση ε, της Νορβηγίας. Έχουμε υπογράψει ένα σύμφωνο με την περιοχή, με την Ορμανδία. Και έτσι γεννήθηκε ο δείκτης της Νορμανδίας. Βασίζεται σε απειλές που εντοπίζονται στην παγκόσμια θετική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και προσμετρούμε την απειλή κατά της ειρήνης για όλες τις χώρες στον κόσμο. Ο δείκτης προετοιμάστηκε από, το, ε, ε, από την υπηρεσία έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα στοιχεία τα έδωσε το Ινστιτούτο Οικονομικών Στοιχείων για την Ειρήνη. Η μελέτη παρουσιάζεται σήμερα με τον τοίχο «Χατογράφηση των απειλών κατά της ειρήνης και της δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο» εισαγωγή στο δείκτη της Νορμανδίας. Το περιγράφει αυτό τα αρχικά πορίσματα θα δώσω το λόγο στον κύριο Τιάν Μπασού Θα λάβετε το λόγο από εκεί ή θα έρθετε εδώ. Ελάτε. As I will have to leave. Επειδή πρέπει να αποχωρήσω, θα ευχαριστήσω τον συνάδελφο που θα συνεχίσει την ασκεί τα καθήκοντα Προέδρου εν τη απουσία μου. Κύριε Μπασό, καλώς ήρθατε στην συνεδρίασή μας. Είναι διευθυντής στο EPRS, είναι υπεύθυνο για τις υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη και θα μας κάνει μια παρουσίαση ε, της μελέτης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ετοίμασα την παρέμβασή μου γαλλικά, αν επιτρέπετε λοιπόν. Χρησιμοποιήσω τη γαλλική, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και την ευκαιρία που μας δίνετε σήμερα να παρουσιάσουμε αυτό τον δίκτυ ειρήνης. Είναι μια δουλειά που πραγματοποίησαμε την Άνοιξη φέτος κατά τη διάρκεια της ε, παύσης των, ε, των διακοπών των ευρωεκλογών και πρώτη φορά στο Διεθνές Φόρουμ για την Ειρήνη ε, που έγινε το Μάιο αναφέρθηκε στον δείκτης. Πολλοί συνάδελφοι εργάστηκαν για αυτού η Μόνικα Νογκά είναι παρούσα, ο Φιλίπ Πασόκ και η Έλανα Λαζάρου και ο Φιλίπ Πασό και συνάδελφοι τη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Εξωτερική Πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ για την συλλογική προσπάθεια που κατεβλήθη, για τη δουλειά που έγινε. Το πρώτο ερώτημα που θέτουμε είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαν στόχο να παίξει πρωταρχικό ρόλο ε, υπέρ της ειρήνης στον κόσμο. Καταρχάς πρέπει να έλθουμε στη βάση του ευρωπαϊκού εγχειρήματο που εδράζεται επί της συμφιλιώσεως των ε, χωρών μας. Το ψήφισμα, των, ε, η επίλυση των διαφορών γίνεται με το κράτος δικαίου, μέσω του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή και εντό των πλαισίων των θεσμικών. Βλέπουμε να διαφαίνονται εκ νέου εντάσει στον κόσμο ε, και να αναδύονται εκ νέου συγκρούσεις, οπότε εδώ μπορεί να παίξει ένα ρόλο παραπάνω η Ευρωπαϊκή Ένωση η βάση της εργασίας μας εδώ σε αυτή την Επιτροπή, η βάση των εργασιών μας των ερευνητικών ήταν η παγκόσμια στρατηγική του 2016. Είναι μια στρατηγική την οποία επεξεργάστηκε η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αλλά που εστερνίστηκαν όλα τα σμικά όργανα, η Στατική Ευρωπαϊκή Ενώσεω ή η Στρατηγική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο στρατηγική είναι ότι προσπαθεί να καλύψει το θέμα της ασφάλειας όχι μόνο από την ε, πλευρά έλλειψη συγκρόσεων, αλλά με ολιστική προσέγγιση, σφαιρική, μέγιστα στοιχεία να ληφθούν υπόψη για σφαιρική προσέγγιση υπέρ της ειρήνης. Οπότε στον εντοπισμό των απειλών βρίσκουμε την παραπληροφόρηση, την αλλαγή του κλίματος, μπορούν να αποτελέσουν απειλές για την ειρήνη. Όπως ε, βλέπετε λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και κάποια χρόνια ε, εδώ και 7 χρόνια πήρε το βραβείο ειρήνη για διεθνή συνεργασία, περιφερειακή συνεργασία το 2012 για, την, για το ρόλο που έπαιξε για την ε, προάσπιση της ειρήνης και στην Ευρώπη και στο παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό είναι μια ευθύνη. Εν συνεχεία ένα άλλο στοιχείο που είναι αποφασιστικό για τη δουλειά μας είναι οι προσδοκίες των πολιτών. Εργαστήκαμε στη Γενική Διεύθυνση επικοινωνία βάσει της προετοιμασία των ευρωεκλογών. Είδαμε ποιε είναι οι προσδοκίε των πολιτών που περιμένουν να κάνει περισσότερα πράγματα η Ευρωπαϊκή Ένωση ή που θεωρούν ότι κάνει ή αν κάνουν αρκετά, αν βλέπουμε τα διάφορα θέματα που προτείνονται, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η προώθηση της δημοκρατίας, το θέμα της μετανάστευσης, η προστασία των εξωτερικών συνόρων, η πολιτική άμυνας και ασφάλειας, η πολιτική ασφάλειας. Εκεί σε αυτούς τους τομείς έχουν μεγάλες προσδοκίες οι Ευρωπαίοι πολίτες για προσπάθειες που θα καταβληθούν και στην Ευρώπη αλλά και στο διεθνές προσκήνιο, το παγκόσμιο προσκήνιο. Είναι κάτι που αναφέρθηκε νομίζω και στη διάσκεψη των προσβευτών που έγινε εδώ και μερικές εβδομάδες. Ε, συζητήθηκε το θέμα των προσδοκιών των πολιτών. Πώς παρουσιάζεται λοιπόν ο, ο δείκτης Βλέπετε στους πίνακες εκεί τους δείκτες, όταν κάνει μια παρουσίαση όσον αφορά τα θέματα ποσοτικά, ε, οι αριθμοί είναι πάντα σημαντικοί που παραπέμπουν στο κείμενο. Βλέπετε υπάρχει και επί χάρτου η μελέτη αλλά και στο διαδίκτυο. Εύκολο να φιλομετρήσετε και να δείτε τα γραφήματα. Υπάρχουν δείκτες και εξήγηση της καταστάσεις που επικρατεί σε κάθε χώρα. Γιατί αναφέρεται δείκτης της Νορμανδίας, εξήγησε ότι παρουσιάστηκε τότε στο φόρουμ στην Νορμανδία Όπως είπε, υπάρχει, αποφασίστηκε μια συνεργασία με τις ε, περιφέρειες, το Κοινοβούλιο με τις περιφέρειες, αποφασίστηκε πριν τρία χρόνια για να συνεργαστούμε κυρίως με αυτή την περιοχή που έχει ισχυρό συμβολισμό με την απόβαση στην Νορμανδία που έγινε και ε, είναι στη βάση της προσπάθειας των χειρίματος του Ευρωπαϊκού η συμφιλίωση και σε αυτή την περιοχή ε, έχουμε και στην ΚΑΝ έχουμε το μνημείο για την ειρήνη και εκεί έχουμε το μνημείο που έχει τους περισσότερους επισκέπτες στη Γαλλία εκτός από βέβαια από την περιοχή του Παρισιού. Γιατί να δημιουργηθεί ο δείκτης σε τι διαφέρει από τους ε, υπάρχοντες δείκτες. Ιδού λοιπόν, η αξία του δείκτη είναι ότι βασίζεται σε 11 κριτήρια που αντλούνται από τη γενική στρατηγική. 11 κριτήρια παρατίθενται τα όπλα μαζικής καταστροφής, η απειλή της τρομοκρατίας, η απειλή από την αλλαγή του κλίματος, η κυβερνοασφάλεια, οι οικονομικές κρίσεις, η ενεργειακή ανασφάλεια, τα έφταστα κράτη, όπως τα αποκαλούμε, το διασυνοριακό έγκλημα, η παραπληροφόρηση, τα fake news και οι βίες συγκρούσεις. Ένα κριτήριο πιο θετικό, η ποιότητα των ε, δημοκρατικών διαδικασιών. Για αυτά τα 11 κριτήρια, σε συνεργασία με το Global Institute for Peace ε, καταρτήσαμε αυτούς τους δίκτες ε, που συναθρίζονται και λαμβάνονται υπόψη σε ένα σφαιρικό δείκτη. Λοιπόν, όσον αφορά την παραπληροφόρηση, για να τα λέμε πιο ξεκάθαρα, δεν έχουμε ε, συγκεκριμένο δείκτη. Βασιστήκαμε στο reporter, στο δημοσιογράφη χωρίς σύνορα, στα κριτήρια αυτά. Και για το διασυνολικό έγκλημα δεν έχουμε κριτήριο, βασιστήκαμε σε ένα δίκτυο που ήδη υπήρχε, που αφορούσε τις ε, ανθρωποκτονίες συνολικά. Βασιστήκαμε σε αυτά τα 12 στοιχεία και αν μπορέσουμε να επιφέρουμε βελτιώσεις θα το κάνουμε στην επόμενη έκδοση του εγγράφου. Λοιπόν, αυτή είναι η γενική προσέγγιση. Δεν αναφερόμαστε μόνο στη φυσική βία, αλλά όλα αυτά που δημιουργούν απειλή για την ανθρώπινη ασφάλεια και βαρύνουν, βαρύνουν σε αυτό το κριτήριο. Αν πάμε στην επόμενη διαφάνεια, βλέπετε ένα χάρτη του κόσμου χρωματιστό, βλέπετε τις χώρες, αυτές που είναι πιο σκούρο χρώμα, είναι αυτές που θερούνται, αυτές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη απειλή. Πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το χάρτη με κάθε επιφύλαξη. Επιφυλακτικά λοιπόν, κοιτάξτε. Δεν αφορά τις συγκρούσεις, τις παρούσες η εικόνα, ούτε τις απειλές που αντιπροσωπεύει μια χώρα για τους γείτονες για τον κόσμο. Αλλά δείχνει πόσο ευάλωτες είναι οι χώρες μέσω ε, βραχυπρόθεσμα, πώς απειλείται η ανθρώπινη ασφάλεια εκεί βάση, ε, με, ένα σύνολο, σε ένα, με βάση ένα σύνολο κριτηρίων. Αυτό το, το, το, το καλάθι των κριτηρίων το αποκαλούμε, θα μιλήσω αγγλικά τώρα, παρουσιάζω τις διαφάνειες και σας καλώ αν έχετε το έγγραφο στο χαρτί να πάτε σελίδα 5 γιατί είναι πιθανότατα πιο εύκολο να το διαβάσετε. Όπως είπα για την παραγωγή των δικτών με το Global Institute for Economics και Greece ε, και Crisis ε, συνεργαστήκαμε για κάθε χώρα, για κάθε διάσταση των 11 κριτηρίων που ανέφερα, μπορούμε να παράγουμε αυτό το διάγραμμα. Μπορούμε να παράγουμε και συγκρίσεις ε, σε περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτό το γράφημα τι βλέπετε. Γίνεται σύγκριση της κατάστασης που κρατεί στην Ευρωπαϊκή χώρα των 28 με τον υπόλοιπο κόσμο. Με γαλάζια βλέπετε την Ευρωπαϊκή Ένωση και με πορτοκαλί τον υπόλοιπο κόσμο. Τι βλέπουμε, ότι η Γενικά Ευρωπαϊκή Ένωση τα πάει καλύτερα όσον αφορά την ευαλωτότητα εν συγκρίση με τον υπόλοιπο κόσμο. Όμως έχουμε και εμείς αδυναμίες, είμαστε και εμείς ευάλωτοι, πιο συγκεκριμένα για την ενεργειακή ασφάλεια, η ενεργειακή ανασφάλεια, είμαστε πιο αδυναμοί από ό,τι οι άλλες περιοχές στον κόσμο. Επίσης, ακόμα και αν είμαστε ε, πιο πάνω, δεν είμαστε ε, τελείως προστατευμένη τον κίνδυνο για την κυβέρνηση ασφάλεια και από την απειλή από την αλλαγή του κλίματος ε, υπάρχουν απειλές. Βλέπετε με αυτό το παράδειγμα πώς άμεσα θα χρησιμοποιήσουμε το δίκτυο, γιατί για κάθε χώρα ή για κάθε περιοχή, για κάθε περιοχή του κόσμου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το διάγραμμα και να δούμε που ε, βρίσκονται τα ισχυρά σημεία και τα δύναμα. Μπορούμε να κάνουμε και συγκρίσεις ε, με μια περιοχή μια ολόκληρη Ήπειρο με τη Λατινική Αμερική να έχουμε μια άποψη σαν πολιτική οργάνωση Μερκοσούρ, χώρες Μερκοσούρ. Να γίνει αυτή η κατάταξη για κάθε περιοχή. Μπορούμε να δούμε ποια είναι η θέση της χώρας εντό τη περιοχής, εδώ στα γραφήματα που βλέπετε. Βλέπετε Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία, ζητώ συγγνώμη, και σε σελίδα 23 στο έντυπο. Βλέπετε ότι έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό φάκελο για Ινδία και την Ισία με εξηγήσει. Γίνεται ποιοτική ανάλυση που συνδέεται με τα διαγράμματα. Τα γραφήματα, διαγράμματα δεν παρουσιάζουν την πλήρη εικόνα, την πραγματικότητα. Υπάρχουν και υβριδικές απειλές, συνδυασμός απειλών. Από τα 11 κριτήρια με άλλα στοιχεία που περιγράφουμε στο κείμενο. Στην ποιοτική ανάλυση για 20 χρόνια χώρες προσπαθούμε να έχουμε μια δειγμολητική παρουσίαση της γειτονίας και της κατάστασης που επικρατεί στις διάφορες υπήρους. Βλέπετε εδώ και θα το είδα και στο χάρτη πριν ότι εξεπλάγημεν από την κατάσταση στην Ινδία βλέπουμε εκεί ότι υπάρχει συσσόρευση απειλών που είναι κάτι ανησυχητικό όσον αφορά αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ας πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε το δίκτυο αυτό. Υποστηρίζει κοινευωστικό έργο, έχει επιρροή, επηρεάζει την επιρροή του Κοινοβουλίου, παρουσιάζει μια εικόνα των απειλών στον κόσμο, που έχει χρησιμοποιηθεί ποικιλό σαν εργαλείο ενημερωτικό μέχρι τώρα δεν είχαμε μηχανισμό αξιολόγηση κοινών απειλών. Τώρα υπάρχει τέτοιο μηχανισμό. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι ένα εργαλείο για έλεγχο. Το Κοινοβούλιο λοιπόν χρειάζεται αυτή την εμπειρογνωμοσύνη και τα στοιχεία ανάλυση, να τα έχει στη διάθεσή του αυτά τα στοιχεία για να μπορεί να ασκήσει το ρόλο του, του ελέγχου. Είχαμε την ακρόαση του είπα του εκπροσώπου και τι περασμένε εβδομάδες είχαμε ακροάσει των υποψηφίων επιτρόπων για ανάπτυξη, για διεύρυνση και γειτονία και σαν και τακτικά γίνονται ακροάσεις των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ενώσης, αλλά είναι καθημερινό εργαλείο για σας, μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε μέσω των εργαλείων που βρίσκονται οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι και μπορεί να γίνονται και διάφορες συγκρίσεις. Θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά το μέλλον του δίκτυ τι μπορούμε να προβλέψουμε και μετά μπορούμε να πάμε σε ερωτήσεις και απαντήσεις. Να πω λοιπόν θα αυτό τον πόνο να το διαθέσουμε στο διαδίκτυο και να υπάρχουν γραφήματα διαδραστικά. Οι χρήστες θα μπορούν να πατάνε το κουμπί πάνω στην ε, χώρα που τους ενδιαφέρει, να έχουν διάφορα καλάθια με στοιχεία προς τη διάθεσή τους και να επιλέγουν ε, ανάλυση των διαφόρων στοιχείων και να έχουμε και επίκαιρα στοιχεία. Έχουμε στοιχεία για το 2019 και θα επικαιροποιηθεί, θα επικαιροποιείται η ιστοσελίδα τακτικά για να βλέπουμε αν αυξάνεται ή μειώνεται ο κίνδυνο. Ελπίζω αυτή η έρευνα να σας είναι χρήσιμη. Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την έκθεση αυτή. Είμαστε διάθεσή σας για συζήτηση για προτάσεις για βελτίωση και συνάδελφοί μου και εγώ, αν χρειάζεστε περαιτέρω ανάλυση για κάποια συγκεκριμένη χώρα, με τα χαράς να σας βοηθήσουμε. Αυτά και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εγώ και οι συνάδελφοι είμαστε έτοιμοι για ερωτήσεις, για σχόλια, για προτάσεις, αν υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, uh, Mr. Μια πολύ γενική ερώτηση δική μου. Η μελέτη έχει πολλά συναρπαστικά στοιχεία και διαγράμματα. Και είπατε ότι χρειάζεστε πιο ποιοτική ανάλυση. Θα συμπληρώσετε λοιπόν αυτή τη μελέτη με πιο ποιοτικά τρισδιάστατα στοιχεία. Ή αυτό το κάνουν άλλοι. Και ο κύριος Πέτρας έχει μια ερώτηση. Ευχαριστώ. Σας συγχαίρω. Καταπληκτική μελέτη. Δύο ερωτήσεις. Για τη μεθοδολογία. Για ορισμένες χώρες τη συγκρίνεται με την περιοχή όπου βρίσκονται. Την Τουρκία τη συνδέεται την, ε, συγκρίνεται με την Ευρώπη για το επίπεδο απειλή. Γιατί ενώ άλλες χώρες τις ε, συγκρίνεται με την ευρύτερη περιοχή τους. Στη σελίδα 5 επίσης μας δίνεται ένα παράδειγμα. Παράδειγμα, ας πούμε, των χαρακτηριστικών ειρήνης, του προφίλ ειρήνης, για να καταλάβουμε πώς ε, λειτουργεί η μεθοδολογία σας. Γι' αυτό μας το δίνετε αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή η Ευρώπη σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι σωστή η παρουσίαση εκεί ή είναι παράδειγμα μεθοδολογίας. Γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η σελίδα 5 μας δίνει μια σαφή εικόνα ε, πώς θα πάει η Ευρώπη σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Και κάθε χώρα μπορεί να συγκριθεί με την Ευρώπη, έτσι δεν είναι. Αφού συγκρίνεται την Τουρκία με την Ευρώπη. Γιατί συγκρίνεται λοιπόν, ξαναλέω, την Τουρκία με την Ευρώπη και τι άλλε χώρε με την ευρύτερη περιοχή του. Παρακαλώ κύριε Μπάσο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Πολύ ενθαρρυντικά. Ναι. Είναι μείζον πρόγραμμα τα ποσοτικά στοιχεία είναι ακόμη τα κυριότερα. Κοιτάξτε, όπως είπα για την Ινδία, υπάρχει ένα αθρηστικό αποτέλεσμα διαφόρων απειλών που μας ανησυχούν. Ο δείκτης λοιπόν είναι σημαντικός, αλλά πρέπει να βλέπουμε πάντα τα αποτελέσματά μας σε ευρύτερο πλαίσιο. Γι' αυτό έχουμε και αυτές τις ε, τα επεξηγηματικά σημειώματα που εξηγούν την βαθμολογία της κάθε χώρας. Θέλουμε να καλύψουμε, αν όχι όλες τις χώρες, πολύ περισσότερες. Και θα είναι στο ίντερνετ. Μπορεί όποιος θέλει να το κοιτάξει. Κοιτάξτε, όχι, είναι ουσιώδη αυτά τα στοιχεία. Πραγματικά, στην ε, σελίδα 5 συγκρίνουμε την κατάσταση των 20 χωρών της Ένωσης με βάση τα στοιχεία που έχουμε με την κατάσταση στον υπόλοιπο κόσμο. Λέω για παράδειγμα ότι από πλευρά ενεργική ασφάλεια δεν τα πάμε όσο ο μέσο όρο του υπόλοιπου κόσμου. Όντω αποδεικνύεται αυτό. Καλό λοιπόν είναι να μπορούμε να δούμε σε ποια σημεία είμαστε ευάλωτοι. Κοιτάξτε, μα η Τουρκία είναι χώρα διεύρυνσης μέχρι στιγμής έτσι δεν είναι. Άρα τη συγκρίνουμε με την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αλλά όταν θα έχετε όλα αυτά τα στοιχεία στο ίντερνετ θα είναι δυνατόν να συγκρίνετε την Τουρκία με το Μερκοσούρ για παράδειγμα. Να παίξετε με τις παραμέτρους. Ο δείκτης είναι ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι εξομοιώσει θέλετε. Κοιτάξτε, αν δείτε τώρα την κατάταξη των χωρών. Η Κωνσταντίνα νομίζω έχει το ίδιο επίπεδο, μέσο επίπεδο απειλών με τη Γεωργία. Λένε πολύ διαφορετικέ οι χώρες. Την κατάσταση πραγματικά σε μια χώρα μπορείτε να την καταλάβετε μόνο αν δείτε αυτό το διάγραμμα για τα 11 διαφορετικά είδη απειλών. Γι' αυτό λοιπόν θα το έχετε προσβάσιμο στο ίντερνετ για να το χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε. Τώρα για τη μεθοδολογία. Στη σελίδα 4 του παραρτήματος έχετε τον πίνακα 1 όπου φαίνεται σαφώς πώς χρησιμοποιούμε τους διάφορους δείκτες. Για παράδειγμα, από πού παίρνουμε στοιχεία για τις οικονομικές κρίσεις από την Παγκόσμια Τράπεζα και για την ε, παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και για άλλους δείκτες από άλλες πηγές. Ξέρω ότι μπορεί κανείς να αφισβητηθεί, μπορεί κανείς να αφισβητήσει τα στοιχεία μας. Γι' αυτό θέλουμε η μεθοδολογία και οι πηγές μας να είναι απόλυτα σαφείς. Επαναλαμβάνω. Γι' αυτό το καλάθι. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την παγκόσμια στρατηγική του 2016 ως σημείο αναφοράς. Γιατί συμφωνήθηκε από τα θεσμικά όργανα. Είναι το σημείο αναφοράς μας για την έρευνά μας. Αλλά ξέρουμε ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η παγκόσμια στρατηγική. Χθε είχαμε την ακρόαση του υποψηφίου αντιπροέδρου και υπάτου εκπροσώπου μπορεί να καταρτήσει μια άλλη στρατηγική, να αναθεωρήσει την τρέχουσα. Οπότε θα προσαρμόσουμε και το καλάθι μας. Αλλά αυτή είναι η βάση μας μέχρι στιγμής. Ωραία. Ο κ. Πίτερς ήθελε να συμπληρώσει. Κοιτάξτε, άμα διαβάζει κανείς, μπερδεύεται λίγο. Το παράδειγμα σας δίνει την εντύπωση ότι αυτό διευκρινίζει πώς πρέπει να κατανοήσουμε το διάγραμμα και δεν είναι ένα υποθετικό παράδειγμα, αλλά η πραγματικότητα. Τώρα το κατάλαβα. Γιατί η Ρωσία, για παράδειγμα, για μένα τουλάχιστον και ίσως και για άλλους, είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουμε τη Ρωσία για την Ευρώπη. Μου είπατε αυτό είναι δυνατόν. Θα μπορείτε να κάνετε συγκρίσεις. Με βάση τα στοιχεία μπορεί κανείς να συγκρίνει τη Ρωσία με την Ευρώπη ή με άλλες χώρες. Εδώ βλέπω συγκρίνεται τη Ρωσία με την Ευρασία. Νομίζω είναι ενδιαφέρον να μπορεί να συγκρίνει κανείς την, ε, την ε, Ρωσία με την Ευρώπη. Ναι, να ρωτήσω και εγώ κάτι συμπροματικό. Τι εκφράζουν αυτές οι τιμές. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες. ενδεχόμενο επεισοδίου μεγάλης ε, διάστασης ή η ανθεκτικότητα ή η απειλή για την ειρήνη σε μια περιοχή. Κεντρικο, κεντροαφρικανική δημοκρατία. Βλέπω ότι η κυβερνοασφάλεια είναι μηδέν. Άρα είναι πολύ αδύναμη. Αλλά η χώρα αυτή κατά πόσο εξαρτάται από ψηφιακέ υποδομέ. Πολύ λίγο. Άρα τι απειλή είναι για την ασφάλεια και την ειρήνη της. Κυρίως η ειρήνη και η ασφάλεια μοιάζει με αυτό το δίκτυο να απειλείται περισσότερο από την κυρονασφάλεια παρά από την απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων. Μα τι πιθανότητα υπάρχει να υπάρξει κάποιο επεισόδιο κυβερνοασφάλειας που να απειλεί την ε, ασφάλεια της χώρας είναι ο συνδυασμός διαφόρων παραγόντων. Ναι. Θα μπορούσαν να σχολιάσουν οι συνάδελφοι για την Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία. Όμως, όπως σας είπα, δεν υπήρχε μέχρι στιγμής στην ακαδημαϊκή κοινότητα τουλάχιστον ένας δείκτης συγκεντρωτικός όχι, διορθώνει ο μιλητή. για το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας, έχουμε λάβει λοιπόν στοιχεία από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, ένα δίκτυο για την κυβερνοασφάλεια που εκείνος εκπονεί. Και πράγματι, με βάση εκείνη την κατάταξη, η Κεντροφρικανική Δημοκρατία βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά. Όταν δεν είχαν διαθέσιμος κάποιος δείκτη στην ακαδημαϊκή κοινότητα χρησιμοποιούσαμε τους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα για παράδειγμα για την ελευθερία του τύπου. Για τον κύριο Πέτερς, πράγματι τώρα που έχετε την έντυπη έκδοση είναι δύσκολο να κάνετε συγκρίσεις πέρα από αυτές που έχουμε ήδη εκτυπώσει στο βιβλίο αυτό, αλλά online θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε μια χώρα και να τη συγκρίνετε με μια άλλη, μια χώρα με μια περιοχή ή μια περιοχή με μια περιοχή. Τώρα, εάν σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα μια συγκεκριμένη σύγκριση, μπορούμε να φροντίσουμε, αν μας το ζητήσετε, να την ετοιμάσουμε για σας. Και αυτό ισχύει και για εσάς και για οποιοδήποτε άλλο μέλος της Επιτροπής μπορεί να ενδιαφέρεται. Ήθελε κάτι να προσθέσει συνάδελφός μου γιατί... για κάποιο θέμα, όχι για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Εκ μέρου και των τριών. Η Έλληνα Λαζάρου είμαι. Μία από τις συνεργάτε που συμμετείχε στη μελέτη. Όσον αφορά τη μεθοδολογία, συμπληρωματικά προ αυτά που είπε ο Ετσιέν, στη σελίδα 5 το διάγραμμα αυτό πρέπει να το δείτε μαζί και με το κείμενο που το συνοδεύει, δεν ξέρω αν προλάβατε, που εξηγεί ότι ως 10 έχουμε τους, το να έχει επιτύχει κανείς τους στόχους του πλήρως και 0 λιγότερο. Ε, και τα χρώματα έχουν σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφού δείτε λοιπόν τον βαθμό και αφού δείτε και το χρώμα που θα σας δώσει τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο για να δείτε συγκεκριμένα από ποιες απειλές έχει προέλθει αυτή η βαθμολογία. Κατά τα άλλα, όπως ελέγχθη, μπορούμε να ε, προσαρμόσουμε, να, να προετοιμάσουμε μάλλον γραφήματα στα οποία να γίνεται σύγκριση οποιασδήποτε χώρες με οποιοδήποτε άλλη, οποιασδήποτε περιοχής με οποιασδήποτε άλλη, και να τα συνδυάσουμε αυτά με οποιαδήποτε επιλογή απειλών. Τώρα για την ανθεκτικότητα, αυτό είναι πράγματι μια δύσκολη έννοια και μας είχε απασχολήσει μιας και είναι μια έννοια που αναφέρεται στην ε, παγκόσμια στρατηγική. Θα δείτε στο παράρτημα τη μεθοδολογία και εκεί καθορίζουμε ε, ποιους δείκτες έχουμε χρησιμοποιήσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε συνδυάσει πολλούς διαφορετικούς δείκτες, δύο-τρεις δείκτες, με κάποιον αλγόριθμο, με κάποιο βάρη. Το οποίο σημαίνει ότι σε ορισμένε περιπτώσεις δεν προσπαθούμε να βαθμονομήσουμε τις απειλέ, αλλά μπορεί να δίνουμε κάποιου πόντου σε μια χώρα εάν έχει προετοιμαστεί για να αντιμετωπίζει συγκεκριμένε απειλέ. Επομένως, ένας δείκτη μπορεί να μην καταδεικνύει μόνο ποιο είναι το επίπεδο τη απειλή που αναμένουμε, αλλά επίσης και το γεγονό ότι κάποια χώρα έχει προετοιμαστεί, έχει δημιουργήσει διαδικασία, έχει ε, την ικανότητα να τις αντιμετωπίσει αυτές τις απειλές. Και βεβαίως αυτά τα μέτρα ε, μπορεί να είναι εξελισσόμενα. Δηλαδή το γεγονό ότι ε, μια χώρα έχει ξεκινήσει πρωτοβουλίε για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή θα τη δώσει κάποιου πόντου, αλλά αυτό θα δώσει τα αποτελέσματα στο μέλλον επανέρχομαι στο ζήτημα της κεντροαφρικανικής δημοκρατίας και του Καναδά σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια. Βλέπετε ο Καναδάς να έχει 9 και η κεντροαφρικανική δημοκρατία 0. Όμως ο Καναδάς ε, Βεβαίω, αξιοποιεί πολύ περισσότερο την πληροφορική γενικότερα, άρα είναι λογικό να είναι και καλύτερη κυβερνοασφάλεια. Επομένω, κατά μία έννοια θα μπορούσε να πει κανεί ότι η κεντροαφρικανική δημοκρατία είναι καλύτερα προστατευμένη, γιατί αν κανεί επιτεθεί στα πληροφοριακά συστήματα του Καναδά, θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά από ότι αν επιτεθεί στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Και ε, είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς πώς περιγράφεται αυτή, αυτό το ευάλωτο ε, με αυτό το δίκτυο, με αυτόν τον αριθμό. Απάντηση. Αν διαβάσετε μια, ε, ε, ένα, μια έκθεση της ΕΣΠΑ με τη συνεργασία των τριών θεσμικών οργάνων αναφέρει ακριβώς αυτό ότι εκείνες οι χώρες οι οποίες είναι λιγότερο διασυνδεμένες με την παγκόσμια υποδομή του ίντερνετ ε, είναι εκείνες που κινδυνεύουν λιγότερο να πληγούν από κάποια κυβερνοεπίθεση, όπως είπατε και εσείς. Ο δείκτης αυτός συμπεριλαμβάνει και αυτά τα στοιχεία. Βεβαίως θα συνεχίσουμε να τον βελτιώνουμε στο μέλλον. Και για να επανέλθω σε αυτό που είπατε ότι χρειάζεται και μια ποιοτική αξιολόγηση. Πέρα από το ότι σκοπεύουμε να κάνουμε περισσότερη ποιοτική αξιολόγηση στο μέλλον, μπορώ να σας πω ότι στην υπηρεσία έρευνας έχουμε και άλλες εκθέσεις ε, για τα διάφορα ζητήματα, στι οποίε μπορεί κανεί να ανατρέξει. Δηλαδή, αν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ζήτημα τη κυβερνοασφάλεια, μπορεί να βρει μια έκθεση τη EPRS για το θέμα αυτό. Επομένω, αν θέλετε, το, ποιοτικ... το συμπλήρωμα με τα ποιοτικά στοιχεία είναι όλε αυτέ οι εκθέσει, όλε αυτέ οι εκδόσεις της EPRS. Ε, Φιλίπ, θέλετε να προσθέσετε κι εσεί κάτι. Σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση έχει σχέση και με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε αυτές τις και, σταθμίζουμε αυτές τις 11 α, απειλές. Εμείς τις έχουμε σταθμίσει ισότιμα. Αλλά βεβαίως αν το σκεφτεί κανείς, η ε, ο κίνδυνος μιας βίας σύγκρουσης είναι πολύ μεγαλύτερος ε, και πολύ μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη στην Αφρική από ό,τι στον Καναδά, ας πούμε. Αλλά ε, επιλέξαμε αυτές τις 11 απειλές επειδή προκύπτουν από την παγκόσμια στρατηγική, του Global Strategy της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν προσπαθήσαμε να δώσουμε εμείς κάποια βάρη, κάποια, να τα σταθμίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Το οποίο σημαίνει ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό να δει κανείς την ποιοτική ανάλυση, τα ποιοτικά στοιχεία, για να μην παραγνωρίσει τη σημασία που μπορεί να έχει μια απειλή ή ένα πρόβλημα για μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή του κόσμου. Mm. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τον κύριο Μπασό και όλους τους συναδέλφους του για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ε, συζήτηση που είχαμε και αυτό το πολύ ενδιαφέρον πληροφοριακό υλικό που μας ε, υπέβαλαν. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τους ε, συναδέλφους, εκτός εάν θα ήθελε κάποιος να θέσει κάποιο θέμα υπό τα διάφορα. Και από ό,τι βλέπω δεν επιθυμεί κανείς. Μπορώ να σας ενημερώσω για την επόμενή μας συνεδρίαση που θα γίνει στις Βρυξέλλες στις 12 Νοεμβρίου από τις 9 μέχρι τις 12.30 και Ολοκληρώθηκε η συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος γενικά ευχαριστεί τους διερμηνείς και εμεί ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Thank